Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin... Καλησπέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την ε, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Έχουμε τι εξή αλλαγέ. Στο σημείο 18, η ψηφοφορία για τι διοργανικέ συνομιλίε σε σχέση με, μια, με ένα κοινό σύστημα θεώρησης διαβατηρίων θα αναβληθεί γιατί δεν έχει καταλήξει ακόμα στις διοργανικές ε, συνομιλίες στο Συμβούλιο. Με αυτή την τροποποίηση προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη κοινό Προέδρου. Γλωσσική, γλωσσική συνδυασμή. Έχουμε όλες τις γλώσσες στη διερμηνία πλην της δανικής, κροατικής και ε, ιρλανδικής Στι κατεξουδότησης συμπράξεις τώρα, 14 Φεβρουαρίου του 2019, έλαβε το σχέδιο κανονισμού 2015-849 το Κοινοβούλιο. Με βάση το άρθρο 55 έχουμε μία περίοδο ενός μηνός με παράταση κατά ένα μήνα για την εξέταση των θεμάτων ε, της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Αν έχετε αντιρρήσει παρακαλώ να τις επισημάνετε. 18 Δεκεμβρίου το Κοινοβουλίο έλαβε δύο κατεξουδότητες συμπράξεις ε, για το ιστορικό ε, ταμείο, ασφαλείας, ταμείο Ασφάλειας και Ταμείο για το Άσυλο, την Μετανάστευση και την Ένταξη. Έχουμε δύο προτάσεις ε, των συντονιστών για δύο προτάσεις από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες με την κυρία Ζήπλος εισηγήτρια για δουλειά μόνο στα αγγλικά των συντονιστών. Προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών 21 Φεβρουαρίου του 2019 στι 2 το απόγευμα, ψηφοφορία 7 Μαρτίου και τελειώνοντας σα επισημαίνω ότι έχουμε αύριο ψηφοφορίε ηλεκτρονικέ στι 11 και 4. Περνώ στο σημείο 3 και την ευκαιρία που μας προσφέρετε τώρα να ακούσουμε παρουσίαση από την Επιτροπή και την, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την κοινή ανακοίνωση του Ιουνίου του 2018 ε, για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των παράνομων πυροβόλων όπλων, νεκρών όπλων, φορητών όπλων, ελαφρού οπλισμού και πυρομαχικών, ασφαλέστερη πλακατοχή για την προστασία των πολιτών και τη σχετική στρατηγική που υιοθετήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2018. Ίσως οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι αυτή η κοινή ανακοίνωση απευθύνονταν στο Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και η ΑΦΕ, την ΤΕΒΕ και η ΙΝΤΑ και έτσι έχουμε προσκαλέσει συναδέλφου από τις τρεις αυτές επιτροπές να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Καλώς ορίζω τους συναδέλφους που είναι παρόντες, κανείς δηλαδή. Πάντως έχουμε καλέσει αρκετούς, θα μπορούσαν να είναι παρόντες. Πρώτη φορά λοιπόν που το Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να εξετάσει και να συζητήσει τα έγγραφα που έχουν κρατηθεί. Έχουμε παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή τα θέματα αυτά για χρόνια και εμείς από τη ΛΥΜΠΕ και οι λοιπές συναρμόδες επιτροπές για τα διτά θέματα το, της ασφάλειας ε, των ε, πυροβόλων όπλων για στα χέρια πολιτών, των μικρών και ελαφρών όπλων. Έχουμε επίσης το ψήφισμα του 12 Δεκεμβρίου 2018 επί τη βάση εκθέσεως της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία και τη θετική ε, εκτίμηση από πλευράς του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της στρατηγικής ε, για τα όπλα αυτά, ε, όπου επισημαίνει το Κοινοβούλιο πως υποστηρίζει την αναθεώρηση της στρατηγικής για την καταπολέμηση των παράνομων πυροβολών όπλων φορετών όπλων και λαφρού οπλισμού λαμβανομένων υπόψη των νέων συνθήκων ως προς την ασφάλεια και την ε, πολιτική ασφάλεια, τεχνολογία κτλ. Και επίσης στο ψήφισμα αυτό, μεταξύ άλλων του Κοινοβούλου, που ε, περιγράφει τα όρια ως προς την αποτελεσματικότητα του κανονισμού 258 του 2012 ως προς την εισαγωγή, εξαγωγή μετάβαση, μεταφορά των ε, μη στρατιωτικού κης χρήσεως ε, πυροβόλων όπλων και μια αυστηρή ε, και επιμελή εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της κοινής θέσεως 2008-944 και πατου Συμβουλίου. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Φλωριανά Σύπαλ επικεφαλής της ε, του σχετικού τμήματος, ε, τμήματάρχη δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Δικαιοσύνης του, και του κυρίου Γιάζεκ Μπούλτσα, ε, κύριου Συμβούλου και ειδικού απεσταλμένου για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Και έτσι θα μας δώσουν τις απόψεις τους από την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ την κυρία Σίπαλα να λάβει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι, που καλέσατε την ε, Κομισιόν και την, ε, ε, και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να σας αναφέρει για αυτή την στρατη... να σας παρουσιάσει αυτή τη στρατηγική που συνδυάζει την προσέγγιση της εσωτερικής ασφάλειας με εξωτερικές πτυχές, με πτυχές της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική αυτή έχει σχεδιαστεί με τρόπο που μας, θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη τη σύνδεση ανάμεσα στο λαθρεμπόριο προβολών όπλων και το οργανωμένο έγκλημα μεταξύ αυτού, μέσα σε αυτό και την τρομοκρατία. Είμαστε πεπισμένοι ότι το λαθρεμπόριο πυροβόλων όπλων είναι απειλή για την ασφάλεια όλων όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορεί να τροφοδοτήσει το έγκλημα, την δρομοκρατία και να διευκολύνει και άλλου τύπου λαθρεμπόριο, όπως για παράδειγμα λαθρεμπόριο ανθρώπων ή τρομοκρατική δράση. Δεν πρόκειται να σας αναφέρω το μακρύ κατάλογο πόλεων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο που έχουν δεχτεί τρομοκρατικές υποθέσεις, ε, επιθέσεις και των οποίων οι πολίτες έχουν απολέσει την ε, ζωή τους κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθέσεων, τρομοκρατικών επιθέσεων με τη χρήση ε, παρόμοιων όπλων. Θέλω να υπογραμμίσω αυτή μου τη σύντομη παρουσίαση ότι η στρατηγική έχει τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, να ενισχύσουμε τον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ε, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, να διευκολύνουμε την συνεργασία και τρίτον, η δέσμευση και επιθυμία να βελτιωθεί η διεθνή συνεργασία. Παίρνοντα τον πρώτο πυλώνα, το νομικό πλαίσιο, το ε, ε, πλαίσιο, οι συνεισηγητές ε, υιοθέτησαν την ε, αναθεωρημένη οδηγία για τα πυροβόλα όπλα το 2017 και αυτή είναι η βάση μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον, το Κοινοβούλιο που βοήθησε στην ολοκλήρωση αυτή της εξέτασης αυτού του θέματος. Μετά την υιοθέτηση της οδηγίας, η Κομισιόν υιοθέτησε ε, μια πράξη κατεξιοδότηση για το σημαντικό θέμα της ε, ανταλλαγή, την προφοριών επί των απορρίψεων ετοιμάτων ε, και ετοιμάζουμε και έναν και υπάρχει και ο κανονισμός του 2012 που αφορά την εισαγωγή, εξαγωγή και ε, ε μετακίνηση ε, ή διάβαση ε, πυροβολών όπλων. Υιοθετήσαμε συστάσεις για να βελτιωθεί η εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή διεξάγουμε και μία ακόμα μελέτη για το πώς εφαρμόζεται. Όλα αυτά για να εντοπίσουμε τις αδυναμίες αλλά ε, και τα δυνατά σημεία αυτού του κανονισμού προκειμένου ενδεχομένως να ε, κάνουμε περισσότερη δουλειά σε αυτό στο μέλλον. Πρόθεσή μας επίσης είναι να είμαστε δραστήριοι στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ένα από τα τρία πρωτόκαλα των συμβάσεων του ΟΗΕ ε, κατά του διασυνορικού εγκλήματος αφορά ακριβώς τα πυροβόλα όπλα. Οπότε ε, είναι ένα πρωτόκολλο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος, συμβαλόμενο μέρος, οπότε αυτή τη στιγμή ε, εξετάζουμε την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Ε, θα, αυτό θα ολοκληρωθεί το Μάρτι στη, το στη Βιέννη και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η διεθνής κοινότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή σε, ε, το, του πρωτοκόλλου αυτού ε, ε, σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Μετά, συνεργασία, επιχειρησιακή συνεργασία. Τα πυροβόλα όπλα είναι προτεραιότητα στο, στον πολιετή κύκλο ε, για το ε, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν, η Ευρωπόλ και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται μαζί και με τρίτες χώρες έτσι ώστε οι αστυνομικέ αρχές ε, των κρατών μελών συνεργάζονται όχι μόνο μέσω ανταλλαγής προφορίων αλλά και με επιχειρήσεις, πραγματικές επιχειρήσεις στο πεδίο. Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή εργασία, η στρατηγική επαναλαμβάνει την ε, προσέγγιση σύμφωνα με την οποία όλα τα κράτη-μέλη απαιτείται να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής των διοκτικών του αρχών προκειμένου να εντοπίζονται τα δίκτυα ε, τα οποία γίνεται λόγος και προκειμένου να γίνονται σε βάθος έρευνες. Τρίτο σημείο της στρατηγικής, τρίτος πυλώνας στρατηγικής είναι η διεθνή συνεργασία. Μιλάμε για ε, διασυνοριακό έγκλημα, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες. Η στρατηγική υπογραμμίζει τα, τη βασική περιοχή ενδιαφέροντος που είναι τα Βαλκάνια, καθώς επίσης Ουκρανία, ε, Λευκορωσία, Μολδαβία, καθώς επίσης και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αυτές είναι οι βασικές περιοχές οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Τρία, δύο σημεία τα οποία θέλω να υπογραμμίσω πριν τελειώσω είναι τα εξή. Πρώτον, Δυτικά Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πρόγραμμα δράσης για τη συνεργασία με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε ε, το πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα δράσης, ενδεχομένως θα χρειαστεί μια καινούργια στρατηγική στο μέλλον. Και δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω, είμαστε δραστήριοι στον διάλογο με όλες αυτές τις ε, χώρες, συμπεριλαμβανομένων και το χρονομένα την Ισία, Λίβανος, Ιορδανία, προκειμένου ε, να ευαισθητοποιήσουμε τους συνομιλητές μας, να εξασφαλίσουμε καλύτερη ψηφιακή συνεργασία ε, να βοηθήσουν να δημιουργήσουν ε, ικανότητες και να δημιουργηθεί, να σχηματιστεί ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπιση των απειλών. Τελειώντας να πω ότι πιστεύουμε πως με αυτή τη στρατηγική αποδεικνύουμε πως η, η μάχη εναντίον των πυροβολών όπλων και των ε, φορητών όπλων θα είναι αποτελεσματική και θα γίνει σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Και τώρα να καλέσω τον κύριο Μπελίτσε να συμπληρώσει αυτά που μας είπε η συναδελφός σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που κάλεσε την ΕΕ να κάνει τις παρατηρήσεις της και να συμμετάσχει στη συζήτηση για τη στρατηγική μας για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων πυροβόλων, μικρών όπλων και ελαφρών όπλων και των πυρομαχικών τους. Θα ευχαριστήσω τους προηγούμενους ομιλητές που βοήθησαν να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική. Είμαστε ικανοποιημένοι που η στρατηγική αυτή, όπως εθετήθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο, αντικατοπτρίζει την διπλή ανακοίνωση της Επιτροπής από τις 13 Ιουνίου. Τη στρατηγική, ουσιαστικά το έγγραφο, ε, εκπροσωπεί και εκφράζει μια συνολική στρατηγική προσέγγιση για την εξωτερική και την εσωτερική μας πολιτική. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην επίσημη και άτυπη συνεργασία μας των Γενικών Διευθύνσεων Home και της ΕΕΔ και πολλών εμπειρογνωμών των κρατών μελών και άλλων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας που κάτσε μια διετία. Πολύ καιρό, αλλά νομίζω δικαιολογημένο από το αποτέλεσμα. Επίσης, να ευχαριστήσω τι προηγούμενες προεδρίε του Συμβουλίου και την τωρινή, τη Ρουμανική, που υποστήριξαν την έγκριση και την εφαρμογή της στατικής. Τα προβλήματα που προκαλούν τα παράνομα πυροβόλα, καθώς και οι απειλές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός, ε, περιγράφησαν ευρέως από την κυρία Σιπάλα. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η στρατηγική δεν έχει να κάνει με το να καταστούν παράνομα τα όπλα και τα πυροβόλα γενικώ, αλλά να μην πέσουν σε λάθο χέρια. Η νέα στρατηγική αντικαθιστά την αντίστοιχη στρατηγική κατά των μικρών πυροβόλων που είχε εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2005. Τον Δεκέμβριο του 2016 προτείναμε να ξεκινήσουμε την αναθεώρησή της με τέσσερι ομάδε παραγόντων υπόψη. Πρώτα απ' όλα τι εξελίξει στον τομέα τη ασφάλεια. Δηλαδή την αυξανόμενη απειλή από την τρομοκρατία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω τι επιθέσει στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν τα, ε, τα ενεργοποιημένα ε, στρατιωτικά όπλα που είχαν ε, εισαχθεί λαχθρέα από τα Βαλκάνια, έπειτα τεχνολογικέ εξελίξεις στα μικρά όπλα και η τεχνολογία παραγωγή του με τη χρήση υπολογιστών ή την ε, τρισδιάστατη εκτύπωση. Έπειτα οι εξελίξεις στον τομέα της νομοθεσίας, όπως η Παγκόσμια Συνθήκη για το εμπόριο των όπλων το Δεκεμβρίου 2014 και τέταρτον οι πολιτικές εξελίξεις, όπως η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εγκαινιάστηκε και άρχισε να τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2015. Η ατζέντα επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση τη διακίνηση των παράνομων όπλων είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε την ειρηνική δικαιοσύνη και ισχυρά θεσμικά όργανα. Να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, υγεία, ισότητα των φύλων και ασφαλή πόλη και κοινότητε. Αυτέ ήταν οι κατευθυντήριε γραμμέ λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική, ε, τη Συνολική Στρατηγική του 2016, για να συνδυάσουμε και την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση των πολιτικών μα. Η αποτελεσματική πρόληψη και η καταπολέμηση της διακριτική απειλής που, που αποτελεί το εμπόριο των πυρομαχικών όπλων αποτελεί τον, τη συνεργασία πολλών φορέων σε διεθνέ, τοπικό και ε, κρατικό επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούν οι τελωνιακοί, οι αστυνομικοί, οι εισαγγελεί, οι συνοριοφύλακε, οι ένοπλε δυνάμει, οι μυστικέ υπηρεσίε, οι διπλωμάτε. Όλοι. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν και στα τρία επίπεδα που προανέφερα. Οι δράσει συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό των προδιαγραφών, την ε, υλοποίηση, την ευαισθητοποίηση, την παρακολούθηση, την επιβολή του νόμου και τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Επίση, λαμβάνουμε υπόψη τον κύκλο ζωή των πυρομαχικών, την παραγωγή του, το εμπόριο, την αποθήκευσή τους και τη χρήση τους, καθώς και την ε, αποκομιδή τους. Εδώ η εξωτερική δράση μας αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, την ε, Ανατολική και Νότια γειτονιά, ε, γειτονία και την Αφρική. Ε, είναι θαύμα που καταφέραμε όλα αυτά τα συμπυκνώσουμε σε 32 σελίδε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ε, πυροβόλων, των μικρών όπλων και των ελαφρών. Συνήθω ε, τα πυροβόλα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των δράσεων των διεκτικών αρχών και τη εσωτερική ασφάλεια. Η οδηγία για τα πυροβόλα, λόγω χάρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δια... κανον... ρυθμίζει τη μεταφορά και την κατοχή των πυροβόλων από... για πολιτικού σκοπού και είναι διαφορετική η χρήση των μικρών όπλων και των ελαφρών για στρατιωτικού κυρίω σκοπού. Αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζοντα όλε αυτέ τι κατηγορίε με μια κοινή στρατηγική, θέλουμε να λάβουμε δράση για όλε τι περιπτώσει. Τώρα μερικέ λεπτομέρειε για τα εργαλεία και ε, τι δυνατότητε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή τη. Εσωτερικώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά ω νομοθέτης. Αυτό το δείχνουν τα πρότυπα για τα απενεργοποιημένα και τα ε, πυροβόλα που έχουν ε, ξαναχρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό ως ε, παράγοντας στην, στις επιχειρήσεις με την υποστήριξη της Europol και της Frontex. Επίσης, ως παροχέας πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως με την βάση δεδομένων COARM, όπου καθημερινά τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταλλάξουν κατάλληλες πληροφορίες και μετά ω χρηματοδότης για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στο Διεθνέ επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά ω ε, ένωση που παρέχει δρομή στι τρίτε χώρε για την αποθήκευσή του, την καταστροφή του πλεονάσματο, την οικοδόμηση δυνατοτήτων, τον έλεγχο των εξαγωγών και ούτω καθεξής. Επίσης, ε, ελέγχει την αποτελεσματική υλοποίηση των πολυμερών συνθήκων και των συμβάσεων, όπως τη συνθήκη για, την, για τον πόλεμο των όπλων και υποστηρίζει και τους διεθνείς οργανισμούς για τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση και τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Επίσης, διευκολύνει τι κοινέ θέσει ε, στα φόρα όπου υπάρχουν συζητήσει σε πολυμερέ επίπεδο. Με θέσει όπως αυτές που αναπτύχθηκαν στις συνεδριάσεις ε, του κανονισμού Βάσεναρ και επίσης ασχολείται με την επιβολή κυρώσεων και τα εμπάργκο όπλων ή οργανώνει ε, πολιτικού χαρακτήρα ή στρατιωτικού αποστολές ε, παγκοσμίω. Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει όλους τους άνωθοι αναφερθέντες ρόλους. Αυτό είναι και ο στόχος της στρατηγικής μας. Να καθοδηγήσουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και εκτός για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη κατοχή όπλων από τρομοκράτες, εγκληματίες και άλλους που δεν έχουν ε, το δικαίωμα και επίσης να ευαισθητοποιήσουμε ως προς την ευθύνη και την υπευθυνότητα για το παράνομο εμπόριο όπλων. Όλα αυτά για να ε, βεβαιωθούμε ότι τα όπλα είναι ασφαλή και προστατεύουμε πραγματικά τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Um, ευχαριστώ συνάδελφοι, έχετε το λόγο εσείς τώρα. Ξεκινούμε με την Birgit. Birgit Σίπερ. Βρε, ευχαριστώ πολύ. Στο συγγνώμη. Έχω παρακολουθήσει κάθε λεπτομέρεια το θέμα. Δεν έχω παρακολουθήσει κάθε λεπτομέρεια το θέμα αυτό, αλλά παρακολουθώντας με προσοχή τις ομιλίες, άκουσα να λέγεται παραλήμενες φορέ ότι χρειάζεται η στρατηγική και ότι υπάρχουν και τεχνικές λεπτομέρειες ε, για την κατασκευή των όπλων που πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, ο κ. Μπρίξ αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν μιλούμε για αποτελέσματα, εννοείται ότι πλέον έχουμε στρατηγική. Ή σημαίνει η λέξη αποτελέσματα πως ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αλλαγές και ως προς τη χρήση όπλων ή την παρουσία τους. Φερρυπίν σε σιτηροδρομικούς σταθμούς κάποιων ευρωπαϊκών πρωτεύουσών. Επίσης, μιλούμε συχνά για ανάπτυξη δυναμικού σε διάφορες χώρες, πολύ καλά. Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής και των νόμων που έχουμε αποφασίσει είναι και η δυνατότητα ήδη να διαγνώσουμε αλλαγέ προς προ την ανάμειξη δυναμικού των κρατών μελών. Γιατί περισσότερη έλεγχη σημαίνει και περισσότερο δυναμικό ελέγχου ε, στα κράτη-μέλη, τεχνικό εξοπλισμό, προσωπικό, εξειδίκευση. Έχουμε δηλαδή κάτι απτό σε αυτούς τους τομείς. Τρίτον, Πιέσει ασκήθηκαν ε, κατά των προτάσεων για τέτοια νομοθεσία λόγω τη εντό εισαγωγικών τρομοκρατία, αλλά αυτό εκφράζει ταυτόχρονα και του φόβου των πολιτών. Και αυτό που βλέπουμε ω συνέχεια που δίδεται σε όλε αυτέ τι συζητήσει είναι πω αυξάνεται η ζήτηση, η απέτηση για νόμιμη κατοχή τέτοιων όπλων. Εδώ δεν βλέπουμε κάποιους κινδύνους, εγώ τουλάχιστον τους βλέπω. Γιατί όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που μπορεί να κατέχουν νόμιμα όπλα, χωρίς όμως τη σχετική κατάρτιση για το εάν, πώς ή πότε μπορεί να τα χρησιμοποιούν. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Μπιργκίτ. Ε, Χερούν, όχι. Θα ήθελα να επισημάνω και προς τους δύο προσκεκλημένους μας ότι αναπόφευκτα, μια και πλησιάζουμε προς το πέρας της θητείας, για διαφόρους λόγους, προφανείς βέβαια, ε, θα λείπουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι. Ευχαριστώ την Πίργκητα για τα ερωτήματά της, όπως και τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες. Ε, ερωτήσεις λοιπόν απευθύνονται και σε εσάς, αν θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι εξ αρχής ανέφερα ότι για μας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε στην Επιτροπή αλλά και σε άλλες επιτροπές στα κράτη-μέλη. Αλλά και ότι προσβλέπουμε και σε περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων στο μέλλον, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και έξω από την αίθουσα και διμερώς, τώρα που μας γνωρίζετε. Ξέρετε σε ποιον θα απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Δικαιοσύνης θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις χωρίς να ισχυρίζομαι πως γνωρίζω τα πάντα και ότι μπορώ να δώσω διεξοδικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σας. Ε, λειτουργικός κύκλος. Ας μην θεωρηθεί δεδομένο ότι στο λειτουργικό κύκλο θα είναι παρόντα τα πυροβόλα. Εμείς έχουμε περιλάβει το θέμα του λάθρεμπορίου στην προσπάθεια αυτή. με την οποία τα κράτη-μέλη αλλά και η υπηρεσία προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις. Και νομίζω ότι αυτό ιδιαίτερα αφορά εκτός από τα κράτη-μέλη και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συνεργασία, να υπάρξει ο κοινό προσδιορισμό των προτεραιοτήτων είτε για διερεύνηση είτε για μια κοινή βάση. Όταν προχωρούμε σε μια συγκεκριμένη δράση για την καταπολέμηση των ε, παράνομα διακινουμένων ε, πυροβόλων όπλων. Αυτό διευκολύνει και την ε, συνεργασία σε επίπεδο Συμβουλίου, τελωνιακών αρχών, διοκτικών αρχών και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μας το ζητούν άλλωστε να το συνεχίσουμε. Και δεύτερον, μπορεί να αυξηθούν τα κράτη-μέλη τα οποία εγκαθιδρύουν εθνικές μονάδες για τα πυροβόλα Και θέλω να επισημάνω ότι χωρί να είναι απαραίτητο οι μονάδε αυτέ να είναι πλήρω ανεπτυγμένε και απολύτω ικανέ μόνε του να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα σχετικό με τα πυροβόλα, είναι απαραίτητο να έχουν τη δυνατότητα τη διασύνδεση, να παίξουν το ρόλο του συνδέσμου. Έτσι αυξάνεται αυτό το δυναμικό στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο και εμεί υποστηρίζουμε και συνεργαζόμαστε και σε οικονομικού όρου, αλλά και σε όρου ανθρωπινών πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μη τι άλλο μπορώ να πω ότι υπάρχει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας με την αστυνομία και η δυνατότητα για την νομοθετική δράση που θα συνδυαστεί με την επιχειρηματική δράση, βέβαια πάντα με την υποστήριξη των κρατών μελών, χάρη στην οποία μπορέσαμε στο παρελθόν, αλλά και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, να δημοσιεύσουμε ε, συγκεκριμένες προσκλήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, για τους φόβους των πολιτών και την τάση που υπάρχει να θεωρεί κανείς ότι αν πάρει όπλο μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τη ζωή και την περιουσία του. Νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το συστήσουμε επί μακρόν. Μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν και τους κινδύνους που φέρνει μια τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχω όμως τίποτα πιο συγκεκριμένο να προτείνω. Αρμοδιότητα για την ε, κατάρτιση των πολιτών και την ε, χρήση των πυροβόλων όπλων μπορεί να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η νομοθεσία σχετική με τους όρους ε, κατοχής, οπλοκατοχής δηλαδή, ή αγοράς πυροβόλων όπλων είναι καθαρά εθνική και σε αυτό δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμπληρώσω και εγώ στην εσωτερική δράση στα όσα συμβαίνουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα αποτελέσματα βεβαίως, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που βλέπουμε από τη στρατηγική αυτή και την εισαγωγή της. Δουλειά γίνεται λοιπόν ως συνέχεια και των προηγουμένων στρατηγικών. Διάφορα θέματα τα οποία έχουμε δει να αναδεικνύονται μετά το 2006 και την υιοθέτηση στο 2005 της προηγούμενης στρατηγικής. Και έτσι όταν έχουμε να κάνουμε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να επισημάνουμε πιστεύω τέσσερα συγκεκριμένες ομάδες αποτελεσμάτων, αφενός με δομέ των πλεοναζών των όπλων και οπλισμών που χρηματοδοτούνται με, μέσα του, της ΚΕΠΑ και αντίστοιχα άλλα χώρες όπως η Λευκορωσία, η Γεωργία, τα Δυτικά Βαλκάνια. Όλα αυτά μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Δεύτερον, έχουμε ενίσχυση της ηλικής ε, ασφάλειας ε, και αποθεμάτων ε, προγράμματα PSSM δηλαδή, έτσι οι αστυνομικέ αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια εξασφαλίζουν και την κατάλληλη κατάρτιση και την προστασία των, των όπλων τους, ώστε να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Τρίτον, ανείχνευση όπλων και πυρομαχικών στις περιοχές συγκρούσεων Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που καταγράφουν όπλα, όπως αυτά ε, κατασχέθηκαν από τρομοκράτες και αναζητούν τις πηγές, την προέλευση των όπλων αυτών και την κοινοποιούν βέβαια στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε αυτά να βελτιώσουν τους μηχανισμούς εξαγωγών όπλων. Και τέταρτον, ε, ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξαγωγές όπλων Παραμένει βέβαια θέμα αρμοδιότητας ε, των κρατών μελών η απόφαση για εξαγωγή όπλων. Ωστόσο υπάρχει κοινή θέση, υπάρχουν κοινά κριτήρια και η δουλειά που κάνουμε τίνει προς την σύγκληση στις πολιτικές για τις εξαγωγές όπλων και ανταλλαγή δεδομένων μέσα, μέσω της ε, βάση δεδομένων που έχουμε, που δημοσιεύουμε εξάλλου και το Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι συμμετέχει ενεργά ε, κάνουμε λοιπόν δημοσιεύσεις ετήσιες για την κατάσταση εξαγωγής όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας, λέει ο Πρόεδρος, για τις παρουσιάσεις σας. Λυπάμαι που δεν υπήρχαν πιο πολλά μέλη της Επιτροπής μας παρόντες. Διακόπτουμε μέχρι τις παρατέταρτο. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Um, and Ας ξαναρχίσουμε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ που δεν το σκάσατε κατά τη διάρκεια της διακοπής. Περάμε στο σημείο 5. Εν σχέση με το λαθρεμπόριο και με την ανάγκη περισσότερων ελέγχων ε, για την προστασία των ε, εργαζομένων, μεταναστών εργαζομένων. Έχει σχέση και με την νόμιμη μετανάστευση. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Θεμελιών Δικαιωμάτων δημοσίευσε μια μελέτη για την εκμετάλλευση, εργασιακή εκμετάλλευση των μετακινούμενων εργαζόμενων, μεταναστών εργαζόμενων συγκεκριμένα, με και μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013. Οι μελέτες που θα παρουσιαστούν σήμερα είναι η συνέχεια αυτής της έρευνας. Η πρώτη αφορά ε, τη φύση και τις α, απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο πρόβλημα της εκμετάλλευσης και το δεύτερο, δεύτερο κομμάτι στις εμπειρίες και τις απόψεις ξένων εργαζομένων. Θα δώσω ε, έδωσαν το λόγο στους, στα θύματα, κάτι που είναι αρκετά πρωτότυπο και ιδιαίτερα για τους ε, εργαζόμενους τρίτων χωρών χωρίς ε, νομοποιητικά έγγραφα. Έχετε κάποια αντίγραφα εδώ αν θέλετε. Θα δώσω το λόγο στην Λουντοβίκα Μπάμφη, Program Management manager ε, κοινωνικής έρευνας για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ε, FRA, την Υπηρεσία Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, μεγάλη χαρά έρχομαι σήμερα εδώ για να μοιραστώ μέσα σας κάποια από τα ευρήματα του της δεύτερη μελέτη μας. Θα ήθελα πριν να δώσω τα αποτελέσματα να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τις προσωπικές ιστορίες που συλλέξαμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν από το Νεπάλ που προσ... να δουλέψει από μια εταιρεία ε, για να κάνει γεωργικές εργασίες στην Πορτογαλία του δώσε ένα συμβόλαιο για 200 ευρώ, λίγα σχετικά το οποίο υπέγραψε γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα, ήταν στα πορτογαλικά, έδωσε και τα στοιχεία τη ταυτότητά του, 300 ευρώ έπαιρνε το μήνα για πάνω από 200 ώρες εργασίας το μήνα με 15 λεπτά διάλειμμα την ημέρα. Ε, κάτι που δεν αναφέρονταν στο πρόγραμμα, στο συμβόλαιο και που μετά ε, ανακάλυψε ήταν ότι είχε και επιβάρυνση από τα 307 ευρώ θέματα για την κοινωνική ασφάλιση άλλα. Και επιπλέον βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, την ε, θέρμανση, ψήξη το καλοκαίρι ε, και με όλες τις δύσκολες συνθήκες έμεινε για να δουλέψει θεωρώντας ότι ε, θα τηρήσει την υπόσχεση του για νομοποίηση ο εργοδότης, κάτι το οποίο θα ήταν δυνατό στην Πορτογαλία και τη συνέχισε να δουλεύει με αυτές τις συνθήκες. Έγινε λοιπόν επιθεώρηση από την επιθεώρηση εργασία, κατά τη διάρκεια τη οποία είπαν ε, οι εργοδότες στον εργαζόμενο αυτό να πει ψέματα για τις συνθήκες εργασίας του και να πει ότι είναι ικανοποιημένο όπως έπραξε. Σε ένα δεύτερο έλεγχο, ο εργοδότης ε, ο ε, επιθεωρητή ζήτησε από τον εργαζόμενο, ζήτησε από τον εργοδότη να φύγει από την ε, ε, συνάντηση αυτή για να μπορέσει να μιλήσει απευθεία με τον εργαζόμενο και εκεί αποκαλύφθηκαν όλα αυτά. Αυτό είναι μια πτυχή λοιπόν που ήθελα να σας γνωστοποιήσω. Τι είναι αυτό που μας απασχολεί λοιπόν. Μιλούμε για βαριές μορφές εκμετάλλευσης συνθήκες εργασίας που αποκλίνουν σοβαρά από τις ε, συνθήκες απασχόλησης και μάλιστα σε όρους που αγγίζουν και το ποινικό παράπτωμα στα κράτη-μέλη, διάφορες μορφές εκμετάλλευσης της ε, εργασίας από την ε, δουλεία μέχρι και πιο ελαφρές μορφές εκμετάλλευσης. Εμείς βέβαια ασχοληθήκαμε μόνο με τις αξιόπινες μορφές εκμετάλλευσης σε ένα διάμεσο στάδιο, αυτό που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ε, δουλεία ή καταναγκαστικά έργα. Υπάρχουν άλλες βαριές μορφές εκμετάλλευσης που περιγράφονται άλλωστε και στην οδηγία για τις κυρώσεις του επιβάλλονται εργοδότες όταν, ε, παραδείγματι, υπάρχει δυσανάλογη διαφορά σε σχέση με τους όρους απασχόλησης ε, των νομότυπων εργαζομένων σε σχέση με το παράνομα διακινούμενου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ εύκολο να διαγνώσει κανείς τις διαφορές τις διάφορες μορφές ε, εκμετάλλευσης. Έγινε λοιπόν η έρευνα. Στην περίοδο 13-15 καταρχάς, όπου εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη, έγιναν 700 συνεντεύξεις με διάφορους επαγγελματίε, εξετάστηκαν οι διάφοροι τομεί της οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν τις παράτυπε αυτές τι μορφέ απασχόληση. Εξετάστηκαν οι συνέπειε και οι προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης με την ενίσχυση του ε, ποινικού νομιμοθετικού πλέγματο. πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα και επιτρέπεται ακόμα η παρονομιαυτή απασχόληση, η εξασφάλιση δυνατότητας να ε, καταγγείλουν αποτελεσματικά οι ε, εργαζόμενοι, η βελτίωση της ενημέρωσης, μηδενική ανοχή κτλ. Στη συνέχεια έγινε και η έρευνα που είχε να κάνει με τους ίδιους τους εργαζομένους, τα θύματα δηλαδή της εκμετάλλευσης, συνεντεύξεις με πάνω από 200 εργαζομένους, ένα τέταρτο ε, ήταν υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΛΥΠΗ ήταν ε, υπήκοοι των τρίτων χωρών. Εκ των οποίων και συνολικά το 1 τρίτο αυτών των εργαζομένων είχαν παράτυπη διαμονή. Άρα κοιτούσαμε να δούμε πώς έφταναν στην εκμετάλλευση αυτή, ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας τους, ε, ποια ήταν τα μέσα που χρησιμοποιούνταν από τον εργοδότη, τι δυνατότητες έβλεπε ο εργαζόμενος, πώς μπορούσε να προσφύγει στη δικαιοσύνη αυτό το κομμάτι της έρευνας έλαβε χώρα στα κράτη-μέλη, το βλέπετε, και βλέπετε χονδρικά τους κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπου εμφανίζεται η εκμετάλλευση της εργασίας, δειγματοληπτικά πάντα στο, ε, στα οικιακά, στην ε, σύτηση και στέγη, οικοδομή, γεωργία, αλλά και ε, μικροκαταστήματα, ε, μικροκομωτήρια ε, πλυντήρια αυτοκινήτων, στεγνοκαθαστήρια κτλ. Και επίσης βλέπετε και τα θύματα, την κατανομή με βάση τον αριθμό του, των ομάδων, των μελών μάλλον σε, κατανεμένες σε ομάδες καθεστώτος, είτε ήταν εποχιακή, είτε ήταν με απόσπαση, είτε ήταν ετούνται στο άσυλο, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, άνθρωποι που είχαν έρθει με τουριστική θεώρηση, ε, νόμιμη διαμονή, Ευρωπαίοι υπήκοοι και το καθεξής. Από τα αποτελέσματα που έχουμε λοιπόν ε, συμπηλήσει βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και ως προς την αμοιβή χαμηλότερη από τον ελάχιστο μισθό ή πολλές φορές δεν δίνονταν να κάνει αμοιβή, προβλήματα σε σχέση με την ε, διαμονή και τη σύντηση, ε, κοινωνική ασφάλιση, υπερορίες, υπεράριθμες μάλλον ώρες, χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπές, χωρίς διάλειμμα δηλαδή και χωρίς διακοπές, Σαββατοκύριακα, Πολλές φορές δεν υπήρχαν συμβάσεις ή εάν υπήρχαν η συμβάση που υπέγραφε ο εργαζόμενος δεν του ήταν κατανοητή γιατί ήταν μόνο στην γλώσσα του κράτους στο οποίο πήγαινε να εργαστεί. Συνθήκες εργασίας, συνθήκες διαβίωσης πολύ κακές. Στο ίμιση βλέπουμε ότι τη στέγη την παρήχε ο εργοδότης σε οικιακούς βοηθούς, για παραδείγματι, ή σε γεωργικές εργασίες, είτε στο σπίτι, είτε στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, με πολύ κακές συνθήκες, όταν παρήχε τη στέγη ο ίδιος ο εργοδότης. Πώς γίνεται όμως η προσέγγιση, πώς καταλήγουν οι ε, εργαζόμενοι αυτή στα, τα δίκτυα. Συνήθως πρόκειται για γνωριμίες που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι για να βρουν μια θέση εργασίας, αλλά υπάρχουν και κάποιοι διαμεσολαβητές. Και εκεί από αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι παρουσιάζουν συστηματικά φαινόμενα ε, βαριάς μορφής εκμετάλλευσης και λαθροδιακίνησης εργαζομένων. Πώς γίνεται αυτό, πώς συμβάλλουν, ε, καταρχάς ε, επιβάλλουν ε, μια αμοιβή για τη διαμεσολάβηση, εκμεταλλεύονται ή λένε ψέματα στον εργαζόμενο έχοντας υποσχεθεί καθεστώς νόμις, διαμονής, διαμονής σε παραδείγματι που δεν υλοποιείται όταν αυτός φτάσει στη χώρα. συμβάσεις ε, διαφορετικές όταν υπογράφονται στη χώρα προελεύσεως και άλλες όταν έχει φτάσει πλέον στη χώρα απασχόλησης ο διακινούμενος, ε, υπεργολαβία, δηλαδή περισσότεροι διαμεσολαβητές αυτή την αλυσίδα ε, απασχόλησης που καθιστούν τα πράγματα ακόμη πιο δυσνόητα για τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο αλλά και για τις αρχές για να αναζητηθεί ποιος είναι ο υπεύθυνο. Από τους εργαζόμενους εμείς Θέλησαμε να μάθουμε τι θεωρούν ω πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ότι ήταν αυτό που μπορεί να του να οδήγησε στην εκμετάλλευση αυτή τη ε, εργασία του, όπω άλλωστε είχε ζητηθεί και στην προηγούμενη έρευνα τρία χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν ο κύριο ε, όρο η κύρια προπόθεση είναι το πόσο ευάλωτοι αισθάνονται στην ε, χώρα όπου παραμένουν εφόσον δεν έχουν νόμιμη διαμονή. Άρα λοιπόν και το ότι είναι παράτυποι και ότι το καθεστώ της διαμονής τους εξαρτάται από την ύπαρξη μιας συμβάσεως καθιστά πιο ευάλωτους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει τι, ότι ε, εάν δεν έχουν νόμιμη, νόμιμα έγγραφα φοβούνται ότι θα απελαθούν, μειώνονται οι δυνατότητες εναλλακτικής αναζήτησης εργασίας, ε, το καθεστώς διαμονής ε, εξαρτάται από την ε, απασχόληση, έχει οδηγήσει σε πολλά προβλήματα επίσης. Ε, παραδείγματι δεν τολμάει ο εργαζόμενος να αναζητήσει έναν άλλον εργοδότη, εφόσον συνδέεται το καθεστώς του από τον εργοδότη του. Ένας άλλος παράγων που έχει ε, διαπιστωθεί ότι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή δεν μπορούν να ενημερωθούν και τα δικαιώματά τους, ότι δεν υπάρχει η επιθεώρηση, η εποπτεία αυτή. Οι επιθεωρήσεις δηλαδή είναι πολύ σημαντικές για την ε, διερεύνηση, για την ανείχνευση της εκμετάλλευσης ε, της εργασίας και βλέπουμε ότι δεν ήταν αρκετά τακτικές, μάλλον ήταν σπάνιες οι επιθεωρήσεις, βλέπετε ανά τομέα δραστηριότητας, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ποτέ δεν ελέγχθηκε ένας εργαζόμενος, γιατί είχαμε ερώτηση και αν ποτέ έγινε κάποια ως έλεγχος, κάποια επιθεώρηση. Επίσης, ε, έχουμε άλλους, άλλους τομείς, όπως στον τομέα των οικιακών βοηθών που μόνο δύο είχαν δηλώσει πως ελέγχθησαν, άλλους τομείς όπου 60% δεν είχαν ε, ελεγχθεί ποτέ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν καθόλου επιθεωρήσεις. Δεύτερον, δεν είναι μη αποτελεσματικές γιατί είναι τεράστιος ο γλωσσικός φραγμός. Άρα για να έχει αποτελεσματικότητα αυτή ο έλεγχος πρέπει να προβλέπεται και παρουσία διερμηνέων ε, και ενό ερωτηματολογίου που μπορεί να είναι κατανοητό και επίσης πολύ συχνά οι αρχές επιθεώρησης έκαναν ε, τις ερωτήσεις τους στον εργαζόμενο παρουσία και του εργοδότη του. Οπότε δεν, υπήρχε το ε, δεν υπήρχαν οι συνθήκες εμπιστοσύνης για να μπορέσει να απαντήσει ειλικρινώς. Μια σειρά από στρατηγικές επίσης των ε, εργοδοτών που στόχο είχαν να υπονομεύσουν τις επιθεωρήσεις αυτές. Είτε υποχρεώναν τον εργαζόμενο να πάει να κρυφτεί όταν ήταν προαναγγελθήσα η επιθεώρηση. Και βέβαια αυτό έχει ένα λόγο η ύπαρξη, η προαναγγελία, δηλαδή να είναι παρόν ο εργοδότη και ο εργαζόμενο. Αλλά από την άλλη, αυτό επέτρεπε στον εργοδότη να στείλει όλου του εργαζόμενου σε ένα μέρο που θα κρυφτούν ή να κατασκευάσει ε, ωράρια εργασίας ε, και καταλόγους εργαζομένων ή να δείξει τον ε, κατάλληλο εξοπλισμό υγείας και ασφάλειας ώστε να ισχυριστεί ότι τηρούνται οι συνθήκες ή και να ασκήσει απειλέ στους εργαζομένους του σε σχέση με τι θα πει κατά τη διάρκεια τη επιθεώρησης. Αυτά συνοπτικά τα παρουσιάζουμε σε μια ειδική έρευνα που αναφέρεται στην ε, αυτοψία στους χώρους εργασίας. Ιδιαίτερα για τους οικιακούς βοηθούς. Επίσης, οικιακοί εργαζόμενοι, οι βοηθοί, βλέπουμε ότι έχουν ιδιαίτερο κίνδυνο εκμετάλλευσης γιατί έχουν μεγάλη εξάρτηση από τον εργοδότη τους ε, καθώς ζουν στο δικό του χώρο, στο χώρο που αυτός του προσφέρει. Εξαρτώνται λοιπόν όχι μόνο για την άδεια διαμονής αλλά και για την διατροφή τους και τη στέγη τους ε, ή από, την, ε, ή από τον εργοδότη επίσης για την θεώρηση διαβατηρίου που λύγει κάθε τόσο έχουν παραδοσιακά ούτως ή άλλως χαμηλότερη προστασία εκεί οι εργαζόμενοι. Υπάρχει επίσης ε, σχεδόν απόλυτη απουσία ε, αυτοψιών από τις αρχές επιθεώρησης εργασίας. Ε, κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση γιατί μένουν μέσα σε ένα σπίτι, δεν έχουν επαφή με άλλους γνωστούς. Επιτοπλίστων είναι γυναίκες, έχουμε να κάνουμε με κινδύνους συναφής με το φύλλο όπως σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλα. και προτάσεις για τα περαιτέρω τώρα. Ε, θα ήταν καταρχάς καλύτερη ρύθμιση των ε, και παρακολούθηση των υπηρεσιών ε, επάνδρωσης, ενίσχυση του εργατικού δικαίου και των συνθήκων υγείας και ασφάλειας, βελτίωση των αυτοψιών, εξασφάλιση των δικαιωμάτων για τους μετανάστες, ενημέρωση των ε, εργαζομένων, των θυμάτων δηλαδή, κυρίως όταν βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης που ε, αυξάνει τον κίνδυνο, ενίσχυση των αυτοψιών και της παρακολούθησης στο χώρο εργασίας, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τις επιθεωρήσεις εργασίας στην αστυνομία και τις λοιπές αρχές, περισσότερες αυτοψίες, αλλά όχι μόνο περισσότερες αριθμητικά. Πρέπει να γίνονται με στρατηγικό τρόπο, να είναι πιο αποτελεσματικές, να προβαίνουν σε μια ανάλυση στρατηγική του κινδύνου και του αποτελέσματος. Δηλαδή να αναζητούν ποιοι είναι οι τομέι ο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο ο εργαζόμενος ανάθεση σε αρμόδια σώματα να προσδιορίσουν και τι σημαίνει εκμετάλλευση της εργασίας και αυτό όχι μόνο σε επιθεωρήσεις εργασίας αλλά και λοιπά σώματα που έχουν αρμοδιότητες ε, και για την υγεία και την ασφάλεια ή τελωνιακές αρμοδιότητες κτλ. Ε, πρέπει να αποφεύγεται η εξάρτηση από τον εργαζόμενο, δηλαδή ε, η άδεια εργασίας να μην συνδέεται αποκλειστικά με έναν εργοδότη, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει προϊστορικό εκμετάλλευσης και καταχρήσεων. Ε, πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν τρόπους ώστε μια άδεια παραμονής εάν λήξει το συμβόλο του εργαζομένου που πρόκειται από τρίτη χώρα να μην ε, έχει σαν άμεση συνέπεια πως εκπνέει και η άδεια διαμονής, ε, να υπάρχει δυνατότητα και για θεωρείς διαβατηρίων ε, ε, επιπλέον και η δυνατότητα βεβαίως να μπορεί να καταγγείλει ο εργαζόμενος σε όρους ασφαλείας προβλήματα σε σχέση με την απασχόλησή του και έτσι ώστε να μην έχουν την προτεραιότητα τα ζητήματα της ε, μετανάστευσης ή της, ε, των μεταναστευτικών αρχών ή παρεμπόδισης μετανάστευσης, αλλά συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η παραθυσίαση. Έχετε ερωτήσεις. Εκεί που ξεχνάω να πω ότι κρίμα, ζητήσω συγγνώμη κλπ. Κάποιος με σώζει πάντοτε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρουσα και με κάποιο τρόπο σοκαριστική. Ε, Μια-δυο ερωτήσεις. Ένα από τα σημεία σας ε, είναι ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι αυτή η μετάσταση είναι παράνομη, παράτυπη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ε, έρθει με, στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών και μετά δεν βρίσκανε δουλειά ή είναι άνθρωποι οι οποίοι, ε, στους χορηγήθηκε εργασία ακόμα από όταν ήταν στη χώρα τους και ήρθαν παράνομα. Μετά, η, η ενδιάμεση είναι εθνικές εταιρείες που λειτουργούν σε κάθε χώρα ή πιο διεθνείς ε, εταιρείε αυτή η ενδιάμεση. Δηλαδή, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε μια χώρα ή σε περισσότερες. Και τρίτον, την περασμένη εβδομάδα έγιναν τελικές διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που έχει στην, ε, μεταξύ των καθηκόντων της και το θέμα ε, της εργασιακής εκμετάλλευσης. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί η FRA με την ε, αρχή αυτή και τα κράτη-μέλη. Το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Γερούν. Μια πιο πλατιά ερώτηση. Ως η υπηρεσία ανθρωπιφάντων θεμελιών δικαιωμάτων, ε, συζητάτε το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης και των ενδεχόμενων μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν. Ε, ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερεύσει. Έχουμε δύο θέματα εδώ. Πρώτον, την υφιστάμενη νομοθεσία περί των εποχιακών εργαζομένων, για παράδειγμα, ε, των ερευνητών, των φοιτητών κλπ αλλά αυτά τα μέτρα είναι θετικά σίγουρα. Μία από αυτές τις οδηγίες ε, ήταν και δική μου έκθεση, αλλά αφορούν πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις. Ε, δεν είμαι σίγουρος καν για το πώς και πόσο εφαρμόζονται. Ε, η Κομισιόν ήταν να εξετάσει το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης με ποσοτικά στοιχεία, δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Δεδομένου όμως ότι στην επόμενη θητεία δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια ισχυρή φωνή υπέρ της νομ... νόμιμης μετανάστευσης, διότι ο κόσμος τη φοβάται. Φοβάται γενικότερα τη μετανάστευση. Οπότε είναι ένα μέτρο, είναι ο μετανάστευση που βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών να δυσκολεύονται να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε εσείς Ρεαλιστικά τώρα. Βλέπετε κάποιο πλεονέκτημα στο να ζητήσετε ή να πιέσετε να ληφθούν μέτρα για την νόμιμη μετανάστευση. Ε, αν δεν υπάρχει καθόλου το θέμα στην ατζέντα, προφανώς δεν θα μπορούσαμε και να νομοθετήσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι. Και δεν θέλω να παρέμβω στο πώς θα ψηφίσουν οι συνάλφοι για το θέμα της μπλε κάρτας που θα έρθει σύντομα. Βλέπω εδώ τη Ρομπέρτα. Αναφέρομαι στη μπλε κάρτα και τι έχω την εντύπωση ότι εμείς εδώ την υποστηρίζουμε, αλλά δεδομένου ότι κανένας δεν θέλει την μετανάστευση. Ε, ήμουν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων την περσμένη εβδομάδα το θέμα αυτό είναι στα χέρια των Υπουργών, είναι στα χέρια των κρατών μελών, αλλά υπάρχει μεγάλος φόβος και κανένας δεν θέλει να ακούει τη λέξη μετανάστευση πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη. Τώρα εγώ εδώ ε, βγάζω λόγο. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα γίνει τίποτα για τα πέντε επόμενα χρόνια για την νόμιμη μετανάστευση. Μετά η Κομισιόν θα κάνει αυτό το fitness check, τον έλεγχο του πώ πηγαίνει ο μετανάστευση και δεν θα έχει τίποτα να ελέγξει. Μπρικετέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν λέτε κανεί δεν θέλει να μιλήσει για την νόμη μετανάστευση, μπορεί να έχετε δίκιο. Από την άλλη μεριά ακούγονται και πολλά ψεύδη και πολύ παραπληροφόρηση κυκλοφορεί γιατί η μετανάστευση συμπεριλαμβάνωμένη και τη μετανάστευση για εργασία συμβαίνει όλου του τελευταίους αιώνε από και προς όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι πολλοί δεν θέλουν να το ακούνε, αλλά είναι αλήθεια. Καλό θα ήταν να μιλάμε με νούμερα λοιπόν και με γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Ο Γερούν είπε προηγουμένως ε, ότι είναι πράγματι σοκαριστικέ μερικέ από τι λεπτομέρειε. συμφωνώ και είναι πολύ καλό που μια μελέτη ενδεχομένω θα ε, ευαισθητοποιήσει λίγο το κοινό. Αυτό που όμω είναι σοκαριστικό πιο πολύ είναι ότι όλα όσα αναφέρονται στην έκθεση αυτή δεν είναι τίποτα καινούριο. Γιατί όλα αυτά τα παρατηρούμε εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες ζούμε τέτοιες καταστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Και φοβούμαι ότι ακόμα και αν συμφωνούσαμε για την μπλε κάρτα, και ελπίζω θα το κάνουμε, δεν λύνει το πρόβλημα γιατί το πρόβλημα βρίσκεται στα κράτη-μέλη, το γνωρίζουν, αλλά δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Γιατί τελικά οι εργοδότες είναι αυτοί που ωφελούνται από τους ε, μετανάστες οι οποίοι δέχονται να εργαστούν για χαμηλές μισθές, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, σε πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης, πολύ κοντά στη δουλεία ή στα καταναλωτικά έργα, απολύτως εξαρτώμενοι από τον εργοδότη και τα κράτη-μέλη δεν θέλουν καθόλου, δεν έχουν καμία ε, βούληση να προστατεύσουν τα θύματα και να αλλάξουν την κατάσταση. Ακόμα και όταν ελέγχουν, όταν επιθεωρούν και εντοπίζουν παράτυπους εργαζόμενους, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα θύματα καταναλωτικής εργασίας μπορεί απλώς να σταλούν πίσω στη χώρα τους και ο εργοδότης να πληρώσει ένα πολύ πολύ μικρό πρόστιμο. Πιστεύετε ότι η μελέτη αυτή θα βοηθήσει να αλλάξει κατάσταση στα κράτη-μέλη. Όχι, αλλά είναι καλό που έχει γίνει, λέει ο πρόεδρος. Ε, πολύ σωστά όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν βούληση να αλλάξουν τα πράγματα. Ε, να πω και το εξής. Όταν κάνατε αυτή την, την μελέτη, είδατε τις επιφυλάξεις των κρατών μελών, φαντάζομαι. Ένας άλλος λόγος για αυτές τις επιφυλάξεις, ή μάλλον μία, ένα άλλο ψεύδος, είναι ότι η μετανάστευση ρίχνει τους μισθούς. Ε, αυτό το υποστηρίζουν όλοι, όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν προέρχεται αυτή, η, αυτός ο σχέσμος μόνο από τη δεξιά. Πολλοί λένε, όλοι λένε ότι η μετανάστευση ρίχνει τους μισθούς. Και γι' αυτό το λόγο ίσως τα κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο ίσως να μην θέλουν να νομοθετήσουν ε, δεν ξέρω αν το εξετάσατε αυτό, αν το έχετε εξετάσει θα έπρεπε, διότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα που χρησιμοποιούν πολλοί και λένε ότι φτηνά χέρια εργασίας ε, πλημμυρίζουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι ψεύδο. η ίδια η μετανάστευση δεν ρίχνει τους μισθούς, ε, αλλά ίσως και αυτό να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα κράτη-μέλη αποφεύγουν να νομοθετήσουν. Και το είδαμε αυτό με, τον, ε, με την οδηγία για τους εποχιακούς εργαζόμενους, ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά των κρατών μελών. Um, first of all, the... που έρχονται οι νόμιμοι εργαζόμενοι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Κάποιοι που ήρθαν στα πλαίσια μιας διαδικασίας ασύλου ε, απορρίφθηκε η αίτησή τους. Πολλοί που έφτασαν νομίμως έγιναν παράτυποι στη συνέχεια για διαφορετικούς λόγους. Μεταξύ άλλων, ε, λόγω υποσχέσεων των εργοδοτών να τακτοποιήσουν, να νομιμοποιήσουν την κατάστασή τους, το καθεστώς τους ή να παρατείνουν την αντιπραμονή τους. Δηλαδή πιάσανε δουλειά Ελπίζοντα ότι θα νομιμοποιηθούν και εντωμεταξύ έγιναν παράτυποι. Αυτό είναι και στρατηγική των εργοδοτών. Κάποιες φορές να παίρνουν παράτυπους για να μπορούν να του εκμεταλλευτούν περισσότερο, όπω βγαίνει συμπέρασμα από τη μελέτη. Και κατά πάσα πιθανότητα και σε σχέση με όσα συμβαίνουν τώρα, θα το δούμε και σε λίγα χρόνια, με την κρίση του ασύλου, όπως έχει ονομαστεί και τις απορρευτήσεις αιτήσει, θα καταλήξουμε να έχουμε όλο ένα και περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις. Λιγότερη προστασία δηλαδή. Για τους οργανισμούς και τα πρακτορία ε, έβρεσης εργασίας. συνήθως έχουν κάποιον συνομιλητή σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ε, που ασχολείται με εργασιακά και τους βοηθάει για την πρόσληψη, για τις προσλήψεις. Υπήρχε ένας μικρός αριθμό ε, περιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά γι' αυτό είναι σημαντικό έλεγχο και παρακολουθήση να γίνεται όχι μόνο στα νέα κράτη-μέλη, αλλά και στα παλιά. Ή μάλλον σε οργανισμού τρίτων χωρών. Μπορεί να έχουν εκεί κάποιον ε, ανταποκριτή, για να το πω έτσι. Και το θέμα είναι η νομοθεσία να επιτρέπει την παρακολούθηση και αλλού. Και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό. Ναι. Για την ε, εκμετάλλευση ε, στο χώρο εργασία είναι σημαντικό που αναφέρεται και αυτό. Καλό θα ήταν να υπάρχουν κοινέ επιθεωρήσεις Είναι σημαντικό. Ιδίω σε αυτή την αλυσίδα υπεργολαβιών, συμβάσεων υπεργολαβίας, ε, είναι σημαντικό ένας που έχει περάσει από κάτι κράτη-μέλη να μπορεί να επιθεωρηθεί. Αλλά και για τους ε, μετανάστες που μπορεί να είναι νόμιμοι είναι σημαντικό. Πάντως ε, με μελέτες αυτού του είδους <clears throat> η δουλειά των επιθεωρητών, των οργανισμών επιθεώρησης ε, καθοδηγούνται από μια μελέτη εντεκτύπου η οποία βασίζεται σε μια σειρά από κριτήρια μεταξύ των οποίων είναι στρατηγικές. Οι στρατηγικές που καταρτίζονται μετά από τέτοιε μελέτε. Ο ρόλο τη ΦΡΑ, λοιπόν, του Οργανισμού για τα Θεμελίδια Δικαιώματα, μπορεί να είναι ακριβώ να κοιτάζει σε ποια κράτη-μέλη ε, μπορεί να συγκεντρώσει στοιχεία για την τακτική επιθεώρηση από ελεγκτέ τη εργασία, βέβαια που θα είναι μικρού αριθμού λόγω των περιορισμένων πόρων. Για την νόμιμη μετανάστευση είναι μια από τις συστάσεις της μελέτες. Τη μελέτη. Να βρούμε κάποια προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση. Να δημιουργηθούν τέτοια προγράμματα ώστε ο κόσμο να έχει ε, δίωδο νόμιμη για να έρθει να δουλέψει, όχι να χρειάζεται να ρισκάρει τη ζωή του. Και για να μην βρίσκεται και σε καθεστώς παρατυπίας, δηλαδή να εξαρτάται από έναν εργοδότη και να είναι ευάλωτος σε πιέσει και τάσει εκμετάλλευση. Δεν έχω πολλά να προστάσω. Σημαντικό θα ήταν να γίνει μια επιμελέτη για τα θέματα αυτά. Για τα νόμιμα συστήματα μετανάστευση που μπορεί να έχουν εκπονήσει τα κράτη-μέλη, υπάρχουν κάποια. Και ένα άλλο θέμα θα ήταν ε, τα προγράμματα νομιμοποίησης. Πιο δύσκολο βέβαια αυτό ακόμα, ξέρω εγώ αυτό που έχει η Ισπανία, θα βελτίωνε την κατάσταση των εργαζομένων για, ειδικά για αυτούς που βρίσκονται επί σειρά ετών ε, σε κάποιο κράτος. Ελπίζω η μελέτη αυτή κάτι να αλλάξει. Δεν είναι μια νέα έρευνα. Ίσως αυτό που είναι καινούριο σε αυτή τη δεύτερη φάση είναι ότι ακούστηκαν για πρώτη φορά οι φωνές των θυμάτων. Γιατί στην έκθεση υπάρχει μια σειρά από συστάσεις που έχουν εκφραστεί από τους ίδιους για το πώς θα μπορούσαν να τους προσφερθούν κάποιες υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες υποστήριξης και μάλιστα είπαν εκεί ότι είναι και ικανοποιημένοι με όσα γίνονται τώρα, ή τι θα πρέπει να κάνουν οι ε, αστυνομικοί, η αστυνομία. Πώ μπορεί να βελτιωθεί ο βαθμό εμπιστοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή των θυμάτων. Και για να κλείσω, όταν κάναμε την έρευνα, όχι, όχι, μα την αλήθεια θέλω να πω. Μιλήσαμε κυρίως με ειδικού και όσους εργάζονται στην πράξη. Το πολιτικό στοιχείο δεν μας απασχόλησε πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι πραγματικά κέρια σημασία ζητήματα. Πολύ σημαντικά. Τώρα έχουν περάσει και στο δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων. Νομίζω η Μπίρ και το Γερούν εξήγησαν και δύο ότι είναι ουσιαστική σημασία και προσπαθούμε να τα εξετάσουμε και εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη δουλειά σας, ε, για τη δουλειά που κάνει ο Οργανισμός Μελιδιών Δικαιωμάτων και σίγουρα θα συνεχίσετε και στην επόμενη θητεία με τον ίδιο τρόπο. Και ευχές και καλή τυχή σε όλους όσοι εργάζονται στον ε, ΦΡΑ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 6. Να παρακαλέσω την Ατεγμίντερ, διευθύντρια. Ε, παρακαλώ, ανεβείτε εδώ. to colleagues, um, thank you very much. So, colleagues, I'm glad to... Και τώρα, καλώς ορίζω αγαπητή συνάδελφη την Πάτεκ Μίντερ, διευθύντρια για τα Ταμεία Μετανάστευση και Ασφαλείας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, που όπως ε, θα θυμάστε έχει τη διαχείριση των ταμείων αυτών. και την αστυνομική συνεργασία, διαχείριση συνόρων, περικλής. Ελπίζαμε να δούμε και την DigiJust, αλλά δεν στείλαν κανέναν, Επομένω μόνο εσείς κυρία Κμίντζερ από την DigiHome. Ενημέρωση. Έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα αυτό για μας στη Λίμπε προετοιμασία του πρώτου προσεχού προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου, διαχείριση κοινή, άμεσα ή έμεσα, που ε, προξενεί κάποιε δυσκολίε και στο Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Πάντως είναι δύσκολο για εμά να παρακολουθήσουμε πώς έγινε η διάθεση των κονδυλίων. Στόχοι λοιπόν τη σημερινή ενημέρωση πρώτα, να ενημερωθεί η Επιτροπή μας το 2019 και προγράμματα των προγραμμάτων του 2019. Και άρα θέλουμε δράσει ειδικέ, δράση συνεργασία με τρίτες χώρες, υλοποίηση από τα κράτη-μέλη και διαχείριση των ταμείων μέχρι τώρα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην Πεάτα και περιμένω και τι ερωτήσει των συναδέλφων όσων ιδιαίτερω ασχολούνται με το το δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπεάτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα, ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σας μιλήσω σήμερα. Θα ήθελα τα πρώτα 10-15 λεπτά να σας δώσω μια επισκόπηση για την υλοποίηση του σχεδίου έχω φέρει και ένα PowerPoint, μια παρουσίαση που δεν θα σας παρουσιάσω διεξοδικά, αλλά πολύ ευχαριστώ μετά αν έχετε ερωτήσει να σώσω πιο πολλές λεπτομέρειες. Ξεκινούμε λοιπόν, όπως είπε και ο Κλόντ, με την επισκόπηση, το τελευταίο κομμάτι, εθνικά προγράμματα, που έδωσαν ε, τους λογαριασμούς τους για το 2018 μόλις τώρα, είχαν την προθεσμία δηλαδή μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, ετήσιοι λογαριασμοί. Μια φορά το χρόνο τα κράτη-μέλη μας στέλνουν το λογαριασμό θα πούμε. Και έτσι έχοντας συλλέξει όλες τις πληρωμές, έχοντας καταρτήσει τον κατάλογο όλων των πληρωμών ε, και έχοντας ε, προβεί και στην επαλήθευσή τους και όταν είναι έτοιμα θεωρώντας ότι μπορούν να δώσουν ε, το εύσημα για τις δαπάνες τους, τα στέλνουν σε εμά για καθάριση και εμείς βέβαια στους επόμενους μήνες θα κάνουμε τις περαιτέρω ε, ερωτήσεις για το τι έγινε, πώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια ή συστάσεις για καλύτερη και πιο νομότυπη χρήση. Μια μικρή καθυστέρηση λοιπόν, το λέμε και jet lag, ε, μετά την υιοθέτηση που αργά φέτο, το πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο, ξεκινάμε δηλαδή με το 2015, τώρα έχουμε φτάσει στο 2018, έχουν πάρει τη σειρά τους, έχουν ρονταριστεί τα προγράμματα και έχουμε να κάνουμε μόνο με υλοποίηση αλλά έχουμε και το προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το 2020 που μπορεί να πάρει μέχρι το 2022 για να κλείσουμε οριστικά το 2023 τα ε, τμήματα που αφορούν το το νομικό πλαίσιο. Στο λέω αυτό γιατί εδώ βλέπετε το μπλε, στο μπλε τα ποσά που έχουμε εδώ στα κράτη-μέλη, που έχουμε κατανήμη μάλλον, άσυλο μετανάστευση, το πρώτο το μεγάλο, στη μέση σύνορα και το τρίτο τα μικρότερα ποσά αστυνομική συνεργασία. Δεν ε, μπορείτε να τα δείτε, φαντάζομαι είναι μικρά, αλλά εδώ βλέπετε τις κατανομές ανά κράτος μέλος, ε, τις δεσμεύσεις στο πορτοκαλί και εδώ είναι τα ποσά του 17 διότι Πρέπει τώρα να μας στείλουν βέβαια τα, τις αιτήσει για τις πληρωμές ε, τα κρατημέλη, αλλά την υλοποίηση και τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων τις ε, στέλνουν μέχρι το Μάρτιο, επομένως έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ως προς την υλοποίηση. Εδώ βλέπετε λοιπόν ε, τις δηλώσεις μέχρι το 17 με το κίτρινο και το πράσινο είναι μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή όλο το 18. Τα τρία ταμεία χωριστά που παρουσιάζουν αύξηση. Συνολικά λοιπόν το πρώτο, η ε, ανάληψη υποχρεώσεων το δεύτερο και οι πληρωμές μέχρι το 2017 στο κίτρινο και ε, αιτήσει για πληρωμέ, γιατί ακόμα δεν έχει ε, ληφθεί η σχετική απόφαση για την καταβόλη των ποσών, για το 2018 στο πράσινο. Ε, η απορρόφηση λοιπόν βελτιώνεται από τα κράτη-μέλη και βλέπετε εδώ ανά κράτος μέλος και αναταμείο και πάλι επαναλαμβάνω θα σας δώσουμε την μελέτη αυτή για να τη δείτε πιο προσεκτικά αλλά πάντως έχουμε τις τάσεις, ε, τα ποσοστά μάλλον απορρόφησης και υλοποίησης, αντίστοιχα κόκκινο και μπλε και βέβαια η υλοποίηση πάντα είναι υψηλότερη στις περιπτώσεις λόγω και της διαφοράς που έχουμε το 17 και το 18 με υψηλότερη απορρόφηση που οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ακόμη στατιστικές για την καταγραφή των ε, ποσοστών απορρόφησης που περιμένουμε ε, των ποσοστών υλοποίηση που περιμένουμε το Μάρτιο, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Ταμείο λοιπόν για τα σύνορα, εδώ και στη συνέχεια πάλι μια ένα αντίστοιχο γράφημα, αστυνομία. Είναι μικρά τα γράμματα, στο συγγνώμη, αλλά θα έχετε, όπως είπα, στη θέση σας τη μελέτη. Τι προτείνει λοιπόν, τι δίνει το Ταμείο, τι δίνει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός στα κράτη-μέλη και τι έχει επιτευχθεί χάρη σε αυτά. Έχουμε τακτική ε, λογοδοσία των κρατών μελών με τις εκθέσεις τους. Ε, 2.185 συνολικά έργα για τη μετανάστευση και την ένταξη, Δύο δις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Κατά μέσο όρο τα έργα διαρκούν ε, περί τους 20 μήνες και κοστίζουν περί τα 500.000, 550.000. Αυτή είναι η συμβολή τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρηματοδότηση 75 έως 90% αναλόγως του έργου. να είναι πιο ακριβό από ό,τι μπορεί να προσφέρει σας συμβολή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας δίνω εδώ παραδείγματα στο κομμάτι που αφορά την κοινωνική ένταξη, στο κίτρινο δηλαδή, έχουμε προσφέρει βοήθεια σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του Ταμείου αυτού ε, από εθνικές, τοπικές ή περιφερειακές στρατηγικές. Και επίσης 160.000 ευάλωτοι, ευάλωτα άτομα ή ε, ασυνόδευτα ανήλικα έχουν λάβει ειδική ενίσχυση χάρη στο Ταμείο. Και πάλι για να σας εξηγήσω τα, ε, ψηφία, τα, τα στοιχεία αυτά. Είναι, τα λέμε fund for fun γιατί με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση δαπανούμε τα κονδύλια αυτά για τους στόχους που προβλέπονται. Επίσης έχουμε επαναπατρισμούς, 77.000 εθελοντικοί επαναπατρισμοί που έχουν χρηματοδοτηθεί, από το Ταμείο 24.000 ε, επανεγκατεστάθησαν με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν ε, εκδηλωθεί. Κάτω δεξιά, στο κίτρινο δηλαδή, έχουμε και τη συμβολή μας στην ε, ε μετεγκατάσταση και νόμιμη είσοδο στην Τουρκία με 30.000 περίπου και πάλι έχουμε ποσά που μας επιτρέπουν να επαναπρογραμματίσουμε και να αναθεωρήσουμε τους στόχους για τους οποίους χρηματοδοτούνται τα έργα αυτά. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε για την ε, θεώρηση διαβατηρίων και για τα ε, σύνορα, τις αντίστοιχες δράσης προστασίας. Έχουμε 600 εκατομμύρια περίπου ως ποσό συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, 1,3 εκατομμύρια αντίστοιχα. Επομένως έχουμε 364 προξενία που είτε δημιουργήθηκαν, τα αναβαθμίστηκαν. Έχουμε κατάρτιση προσωπικού γύρου στις 9.000 στη διαχείριση των συνόρων, πάλι χάρη στο ταμείο αυτό. Μετά στο ESF Πολύς Αστυνομίας έχουμε 720.000, μέσο κόστος 387 εκατομμύρια και πολύ άριθμα σχέδια. Εδώ έχουμε τα στιγμιότυπα που δημοσιεύονται. Μία μόνο εικόνα σας δείχνουμε εδώ σαν παράδειγμα. Κέντρο ενσωμάτωση στην κοινότητα στο Βίλνιους, όπου οι ε, άλλοδοποί έρχονται σε επαφή με τους ε, ντόπιου που τους δείχνουν και τις συνθήκες διαβίωσης ε, και τους βοηθούν να μάθουν τη γλώσσα κτλ. Έχουμε ακόμα να ολοκληρώσουμε προγράμματα για το επόμενο διάστημα. Νομική βάση, παραδείγματι, που χρειάζεται ακόμη να ολοκληρωθεί για το ESF και την, ε, τα σύνορα και τη θεώρηση. Εσείς ως αρχή αρμόδια για τον προπολογισμό μας μας έχετε προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση που αναδιανέμεται στα κράτη-μέλη στην προσπάθεια να τα στηρίξουμε για να εντοπίσουν κενά από την αξιολόγηση σέγγενη, από την ε, αξιολόγηση ευάλωτων προσώπων ή για την αγορά εξοπλισμού που θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων για τις ανάγκες τους. Επιπλέον ποσά για την ενσωμάτωση και τους επαναπατρισμούς που επίσης έχετε προσφέρει και ειδικά για το Ταμείο για τα Σύνορα έχουμε κάλυψη στοιχείων του Σέγγεν που για λόγους διαδικαστικούς έρχονται με καθυστέρηση και αναδιανέμονται πάλι στα κρατη με την κλίδα ανακατονομής που προσδιορίζεται στην αρχή της προγραμματικής περίοδου και με αυτή θα κλείσω γιατί είναι ένα δίδαγμα που έχουμε αποκομίσει ότι δηλαδή δεν έχουμε στη χώρα εκεί όπου θα χρειάζονται τα χρήματα ε, τη διαθεσιμότητά τους και άρα κάτι που μπορούμε να εξασφαλίσουμε σαν βελτίωση είναι να καλύπτονται οι ανάγκες είτε από τα εθνικά προγράμματα είτε από λοιπούς διάβλους και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε και στην υποδοχή και στη διαχείριση των συνόρων στις ανάγκες αυτές στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής αλλά και όπου υπάρχουν καθυστερήσεις ε, σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις για την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου και ε, ο προσδιορισμός των εθνικών προγραμμάτων. Τώρα έχουμε μια τελική φάση για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που κλείνει, όπως είπα, του χρόνου. Και βεβαίω πρέπει πια, μια και έχει αρχίσει η συζήτηση για το πολίτε νοσονομικό πλαίσιο, να καταθέσουμε τι νέε προτάσει μα. Τι επεξεργαζόμαστε ήδη. Ελπίζουμε να μην οδηγηθούμε πάλι σε καθυστερήσει στην εφαρμογή. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται πια από εμά. Άμεση διαχείριση. Κοινοτικέ δράσεις και στα δύο ταμεία. ΆΜΕΦ και ΑΕΣΕΦ δραστηριότητε άμεσης διαχείρισης που σημαίνουν τι, ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λαμβάνουμε τις ε, προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, και για εκτέλεση με τις ε, δράσεις, ενωσιακές δράσεις όπως τις λέμε όχι αποκλειστικά δηλαδή για κάποιο κράτος μέλος, αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέσσερα συνολικά έργα τα οποία προχωρούν με τη μορφή το σύμπραξης και αποβαίνουν σε όφελος ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε αύξηση του προπολογισμού με αποκορύφωμα το 2017. Το 2019 το βλέπετε κάπως μειωμένο, τον προπολογισμό, αλλά πάλι είναι υψηλός. Παραδείγματα πολλά έχω να σας δώσω, πολύ σύντομα. Στο ΑΜΕΦ έχουμε 145 έργα που τρέχουν ακόμα. Έχουν να κάνουν με την υποστήριξη στην κοινωνική ένταξη, εκστρατείε ενημέρωση τρίτες τρίτε χώρε, υποστήριξη δικτύων, παραδείγματι, ε, κούσου επαναπατρισμού, δίκτυα επανένταξης ε, που τρέχουν διάφορα κράτη-μέλη, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για μια εναρμονισμένη προσέγγιση στους εκούσους επαναπατρισμούς, περιφερειακή ανάπτυξη των προγραμμάτων ε, προστασίας από το υπατή Αρμοστία και τα λοιπά και αφορούν συγκεκριμένα το κέρας Αφρική ή τη Βόρεια Αφρική με το σύστημα καταγραφής μετά την ε, αποβίβαση και ενημέρωση και συνεργασία με τις χώρες αυτές, αλλά και το καταπίστευμα. Ποσά δηλαδή που πάνε στο καταπίστευμα. Επίσης έχουμε τον πολύ ψηλό αριθμό, τον πιο ψηλό αριθμό έργων στο Ταμείο για την Ασφάλεια και την Αστυνομία. με τους στόχους που έχουν να κάνουν με τα δίκτυα αστυνομικής συνεργασίας, την καταπολέμηση του εργανομένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος. Έχουμε μια γενική πρόταση που ονομάζεται Protect και έχει πολλά ε, στοιχεία περιβολάβει, ιδιαίτερα ασφάλεια των αστικών κέντρων και ιδέες με παραδείγματα για την ε, αποτροπή του κινδύνου για τους ήπιους στόχους θέματα τα οποία ενδιαφέρουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Στον τομέα της αστυνομική δράση επίση έχουμε διάφορους τομείς εντοπίσει μεταξύ των κρατών μελών συνεργασίας. Κύριο θέμα ριζοσπαστικοποίηση και ευαισθητοποίηση και τα σχετικά δίκτυα. Αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών που εξετάζει εναλλακτικέ μεθόδους για την αποτροπή του κινδύνου να ριζοσπαστικοποιηθούν κυρίως οι νέοι κοινωνία των πολιτών και πρόγραμμα ενδυνάμωσης της, ε, αξιόπιστες δηλαδή εναλλακτικέ ε, και αφήγημα αξιόπιστο και πίστικο κατά της τρομοκρατικής προπαγάνδας στα σύνορα ε, μικρότερα προγράμματα και διαχείριση του μικρότερου τμήματος του Ταμείου με εννέα έργα μόνο στόχο έχουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Eurosur μελη ξέρετε εσείς τι είναι Eurosur. Συνεργασία λοιπόν μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, χρηματοδότηση έργων στη Βαλτική, για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων και έχουμε και μια ανοιχτή προκήρυξη για 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, υποστήριξη του μηχανισμού αξιολόγησης της Schengen και ε, θεώρηση. Και τέλος έχουμε την ε, ε αρρωγή σε κατάσταση ανάγκης με τα τρία ταμεία και τα ποσά τους και τον προπολογισμό που ένα 1,4 θα δείτε δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, ένα δις 70.000 εκατομμύρια δηλαδή για το ΆΜΙΦ, από το οποίο 68 εκατομμύρια έχουν ήδη χορηγηθεί για, τα, για την αστυνομία και τα σύνορα και μετά βλέπετε που βαίνει αυτή η άρρωγη συγκράταση ανάγκης. Πάλι είναι πολύ μικρογραμμένα. Το μεγάλο κομμάτι στα αριστερά είναι η Ελλάς και λοιποί παράγοντες, η ε, Πατία Αρμοστία, ε, Οργανισμός για τη Μετανάστευση και άλλοι διεθνείς φορείς που προσφέρουν τη βοήθεια τους στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση μεταναστευτικής ε, κρίσης. Ενώ στο κομμάτι που αφορά τα σύνορα και την αστυνομία είναι πιο ισότιμη η κατανομή πάλι βέβαια με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Βουλγαρία ε, στα μεγαλύτερα κομμάτια που βλέπετε. Έτσι λοιπόν με, αυτές τις, ε, με αυτά γραφήματα βλέπετε ότι μεγάλη βοήθεια παίρνει η Ελλάδα, συνθήκες ε, υποδοχής, διαμονής, προστασίας ανελίκων, διερμηνίας, διαμονής, ακόμη και ξενοδοχεία, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Στην Ιταλία έχουμε επίσης βοηθήσει και για ε, εθελοντικούς επαναστατρισμούς, ε, μέτρα προστασίας, ε, υγεία, προστασία θυμάτων διακίνησης, το ίδιο και για την Ισπανία πρώτες αφήξεις κτλ. Και αυτές οι συνθήκες αφορούν και έκτακτες ανάγκες αλλά και για την Ελλάδα ειδικά την μεγάλη πίεση στα σύνορα Άρα δεν αφορούν όλα τα κράτη-μέλη, μόνο τα, τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής. Για να κλείσω διδάγματα, είναι προσθεμένη αξία τα ταμεία αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν όμως αρκετή ευελιξία και ένας από που τους λόγου του τους οποίους πρέπει να προσφέρουμε έκτακτη βοήθεια στα κράτη-μέλη είναι ότι δεν μπορούμε να διανύμουμε επιπλέον κονδύλια με βάση τι ανάγκε. Δηλαδή πρέπει πάντα να ακολουθούμε την κλίδα κατανομή, όπω αυτή προσδιορίστηκε με στατιστικέ που ανάγονται στο 2008. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κατάσταση το 2008 ήταν πολύ διαφορετική άρα τον κόσμο ε, σε σχέση με αυτή που έχουμε το 2019 και άρα οπωσδήποτε πρέπει σε αυτό να δοθούν κάποιε απαντήσει ε, στο προσχέσιο πολιτέ στο πλαίσιο. Έχουμε συνεργατικέ δράσει με άλλα ταμεία, χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια όπω άλλωστε το έχουμε πράξει και στην, και στην πρότασή μα για το πρώτο τεχές πολιτές στο πλαίσιο. Ε, χρειάζεται απλούστευση γενικά στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τον τρόπο διάθεση των κονδυλίων. Και βεβαίω συντονισμό, περιφερειακέ πολιτικέ, κοινωνικέ πολιτικέ κτλ. Διάφοροι τομεί δηλαδή, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ε, αξιολόγηση άργησε κάπω. Ε, πρέπει να ξεκινήσουμε δηλαδή στην προσεχή περίοδο πιο γρήγορη. Και τελευταία πρόταση, εδώ τελευταία διαφάνεια για την επόμενη περίοδο προτείνουμε κονδύλια να δεσμεύονται μόνο κατά 50% με τις που υποχρεώσεων και το 50% να διατηρείται με την ε, με τη λεγόμενη θεματική διευκόλυνση, δηλαδή με βάση τα προγράμματα εργασίας ε, να προστίθενται επιπλέον ποσά και να διατίθενται επιπλέον ποσά στα κράτη-μέλη ανάλογα με την πρόοδο που έχουν επιδείξει και να υπάρχει και ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να προκύπτει μετά από μια πρώτη ή μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, ένα 10%. Δηλαδή ευχαριστώ πολύ στο σύνολο που μακρηγόρησα και πολύ ευχαριστώ να πάτε στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκμέντερ για αυτή τη διεξοδική παρουσίαση. Ένα μέλο μέχρι τώρα, ο κύριο Λόπε Αγγιλάρ έχει ζητήσει το λόγο, αλλά αν κάποιος άλλος έχει ερώτηση, παρακαλώ μην διστάσετε να το πείτε. Η κυρία Σέπελ χρειάστηκε να φύγει, θα χρειαστεί να φύγει δυστυχώ. αλλά Χουάν. Ευχαριστούμε πάντα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά αυτές τις πλήρεις ε, και καταπιστικές παρουσιάσεις. Μία ερώτηση για τους τέσσερις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Όχι, του περασμένου έτους, του 2018. Τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2018 οι διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και η πατιαρμοστία του για τους πρόσφυγες ε, αναφέρουν ότι έγιναν περισσότερες επιστροφές από ότι αφήξεις παράτυπων μεταναστών. Αυτό είναι εξαιρετική σημασία. Γιατί επανειλημμένως έχουμε αναφερθεί στην διαφορά ανάμεσα στα γεγονότα και τις ε, αντιλήψεις. Ψευδείς πολλές φορές. Ο κόσμος νομίζει ότι η μετανάστευση είναι εκτός ελέγχου, ότι μας κυριεύουν εξαιτίας βέβαια του γεγονότος ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρόχειρη. Τα γεγονότα όμως, τα δεδομένα, δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Πρώτον, η μετανάστευση δεν είναι εκτός ελέγχου. Δεν οφείλεται στα... στον κόσμο αυτό, οφείλεται στα κράτη-μέλη που πολλές φορές δεν συμμορφώνονται καν με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Το γεγονό όμω είναι το εξή. Εξακολουθεί να είναι αλήθεια ε, ότι η, ακόμα και σήμερα οι επιστροφές, οι, οι εθελούσιες επιστροφές και οι μη εθελούσιες επιστροφές, όλες οι επιστροφές μαζί υπερβαίνουν τον αριθμό των αφήξεων παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Χουάν. Δεν βλέπω κανέναν άλλο το λόγο. Να προσθέσω κι εγώ μια ερώτηση. Να δω αν μπορείτε να την απαντήσετε, εν πάση περιπτώσει. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές, έχετε κάποιες πληροφορίες για το προς ποιες χώρες επιστρέφουμε το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών. Επίσης αναφέρατε συνεισφορές στο ε, καταπίστευμα για την Αφρική. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις για αυτό το καταπίστευμα. Όταν εσείς από το Άμιφ ε, συνεισφέρετε, χρηματοδοτείτε το καταπίστευμα, γνωρίζετε σε ποιο, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα. Καταρχήν να απαντήσω την τελευταία ε, ερώτηση, γιατί είναι το μόνο δημοσιονομικό ερώτημα. Πράγματι συνεισφέρουμε, αλλά δεν παρακολουθούμε πού χρησιμοποιούνται αυτά τα ποσά, ακριβώς γιατί μπαίνουν μέσα σε ένα συνολικότερο ταμείο. Όμως η Κομισιόν ε, παρακολουθεί το καταπίστευμα μέσω της ε, Μόνιμης Επιτροπής Διαχείρισης, της Steering Committee. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επιστροφών και το κατά πόσον υπερβαίνουν ω αριθμό τον αριθμό των αφήξεων, πρέπει να το δω. Πρέπει να το εξετάσω. Ε, πού επιστρέφουμε πιο πολλούς είναι ένα μείγμα και πάλι θα πρέπει να ρωτήσω τους συναδέλφους που επιστρεφουμε πιο πολλού, ειναι ενα μειγμα και παλι θα πρεπει να ρωτησω τους αδελφους που εχουν αναλαβει τα στατιστικά. Τα έχουμε τα στατιστικά, απλά δεν τα έχω μαζί μου γιατί εγώ πιο πολύ ασχολήθηκα με τα δημοσιονομικά, τα οικονομικά στοιχεία. Δυστυχώ δεν έχω αυτά τα, αυτές τις απαντήσεις. Πρόεδρος, ε, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τόσο, των τόσο περίπλοκων ζητημάτων. Κάπου πρέπει να εστιάσει η συζήτηση κάθε φορά. Να προσθέσω άλλη μια ερώτηση. Πιο δημοσιονομική. Ε, στις χώρες προέλευσης η ε, κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα κατά πολύ μάλιστα. Αναφερθήκατε και την στήριξη της εθελούσιας επιστροφής και της βοήθειας συνδρομής που δίνουν στους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια καινούρια ζωή στη χώρα τους. Πώς ακριβώς βοηθάτε τους ανθρώπους να βρουν ένα καινούριο, μια καινούργια αιστεία στη χώρα τους, ένα καινούριο σπίτι. Πώς τους βοηθάτε ακριβώς, ε, τους βοηθάτε να βρουν θέσεις, εργασίας, απασχόληση. Μήπως ε, στηρίζεται την περιοχή στην οποία επιστρέφουν. Ε, μέσω του Παγκόσμιου Μεταναστεύσεων ε, βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους διότι ε, ο OIM έχει ένα πακέτο στο οποίο συνεισφέρουμε. Αυτό το πακέτο δίνει ένα χαρτζιλίκι ας πούμε, στους ανθρώπους αυτούς που επιστρέφουν, ένα καταποκοπή ποσό και κάποιο τύπου βοήθεια προκειμένου να ξαναενταχθούν στη, στην κοινωνία και να βρουν δουλειά. Δεν ξέρω βέβαια τελικά αν βοηθούνται, αν βρίσκουν δουλειά για παράδειγμα, αλλά πάντως εμείς συνεισφέρουμε στο πακέτο ένταξης του Παγκόσμιου Οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Αυτά προς το παρόν. Προφανώς όταν δαπανούμε ποσά θέλουμε να ξέρουμε πώς δαπανώνται. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις προφορίες που μας δώσατε. Okay, so now we are... Φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. I'm just Το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης προβλέπει την παρουσία της κυρίας Ιντβέλτ και μια αντιπροσωπεία της Κομισιόν. Μια και είναι εδώ και οι δύο, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση προς αυτή απάντηση προς την Κομισιόν από τις 6 Νοεμβρίου 2018 για το πρόγραμμα iBorder Control από τη Σοφία Ιντβέλτ. Η προθεσμία για την απάντηση της ερώτησης αυτής από την Κομισιόν έχει ήδη περάσει χωρίς να λάβουμε απάντηση. Υπό αυτές τις συνθήκες ο... η κυρία Ιντβέλτ, όπως δικαιούται, ζήτησε το θέμα αυτό να τοποθετεί στην μεσία διάταξη της συνεδρίας σύμφωνα με τον κανόνα 130 παραγραφος 4. Εν τω μεταξύ όμως η Κομισιόν απάντησε στην ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, η συγγραφέας η υποβάλλουσα την ερώτηση θέλησε να παραμείνει το θέμα στην ημερησία διάταξη για να συζητηθεί. κυρία Ιντφέλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι λάβαμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η... στη μακρά μου εμπειρία η Κομισιόν έχει δύο τύπους απαντήσεων. Πρώτον, παρακολουθούμε την κατάσταση. Δεύτερον, ε, δεν ότι δεν τίθεται θέμα. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρα. Η δεύτερη. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα του πώς επίμαχες προτάσεις υποβάλλονται με τη μορφή ερευνητικών σχεδίων. Συνήθως αυτό αφορά την έρευνα της μεταφορές. Αυτά όμως είναι μετρά τα οποία θα έπρεπε να περάσουν από την Επιτροπή μας. Εσείς βέβαια είστε όλοι εδώ, οπότε δεν θα πρέπει να απευθύνομαι σε εσά, αλλά όλα αυτά που διαβάζουμε είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μας μιλούν για το νομικό πλαίσιο του, ελέγχου των συνόρων, του ηλεκτρονικού ελέγχου συνόρων, του, συγγνώμη, του High Border Control. Ε, πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο μηχανισμό ε, ανείχνευσης. Ανείχνευσης ψεύδους κατά βάση ανοιχνευτεί ψεύδους για τέτοιο, γι' αυτό μιλάει. Θα πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και θα βλέπει αν λες αλήθεια ψέματα για να σε αφήσουν να μπει ή όχι από τα σύνορα. Μάλιστα η Κομισιόν λέει ότι το σύστημα αυτό θα συνδέεται και με άλλα συστήματα ελέγχου των σύνορων στο πλαίσιο τη διαλειτουργικότητας. <laughs> Το πολύ αγαπημένο μου θέμα όπω ξέρετε. Επίσης θέλουν τα δεδομένα αυτά τα οποία θα λαμβάνονται από τον ε, ανιχνευτή ψεύδους να ματσάρονται με ε, προηγούμενα ταξίδια. Και, και θέλουν και ένα σύστημα ανταμοιβή με βάση τον αριθμό των επιτυχών εισόδων διαλέψεων συνόρων και τον αριθμό των ε, περιόδων διαμονής χωρίς επεισόδιο. Δηλαδή όσο πιο καλός είσαι τόσο πιο πολλούς πόντους θα παίρνεις. Κινούμαστε προς την κινέζικη κατεύθυνση. Ε, μου φαίνεται σαν πρωταπρολιάτικο αστείο. Δηλαδή θα ξοδέψουμε και λεφτά σε αυτό. Ε, και βέβαια το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται είναι πολύ ε, εύθραυστο. Λέει ότι θα διευκολύνει την πιο ταχεία διάλευση νόρων στα αεροδρόμια. Αστείο. Αν δείτε πόσες, πολλές πόσες πολλές προτάσεις έχουν δικαιολογηθεί με βάση αυτή την αιτιολογία, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Θα ήθελα να ήξερα, έχουν μικρύνει ουρές στα αεροδρόμια τα τελευταία 15 χρόνια με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Και μια-δυο ακόμα παρατηρήσεις. Πρώτον, η Κομισιόν ε, δοκιμάζει αυτό το σύστημα σε μερικές χώρες όπως η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Όχι χωρίς προβλήματα, όχι ανέφελα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λέει, εξέτασαν ένα τέτοιο σύστημα και θεώρησαν ότι είναι υπερβολικό. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ε, δεοντολογικής εξέτασης αυτών των προτάσεων. Δεν είναι τεχνικά ζητήματα αυτά. Η Κομισιόν τα παρουσιάζει ως τεχνικά θέματα, αλλά έχουν ισχυρή δεοντολογική και ηθική διάσταση. Δεν θα τα αποφασίσουν αυτά τα πράγματα οι υπάλληλοι, οι γραφειοκράτες. Είναι πολιτικά ζητήματα και θα πρέπει να συζητώνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά δεν μπορούμε να τη θέσουμε και σε όλους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας και ας ακούσουμε αρχικά την Επιτροπή και την απάντησή τους για ε, την ερώτησή σας σε κάποια σχόλια, Γιώργος Επισόφη. Με συγχωρείτε, αλλά έχω και εγώ παρόμοιε ερωτήσει, Αν γίνεται να τι θέσω ταυτόχρονα, ε, για να λάβουμε μια κοινή απάντηση με τη Σόφη, εάν δεν σα πειράζει. Ωραία λοιπόν, να ακούσουμε την ερώτηση προηγουμένως. Λοιπόν, όταν η κυρία Ίνβελτ έστειλε τι ερωτήσει στις 6 Νοεμβρίου, εγώ στι 7 Νοεμβρίου έστειλα την 00539 ε, 18 και αυτέ δεν έχουν απαντηθεί. σύντομε ερωτήσει. Σε τι επιστημονικά δεδομένα βασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πολιτικό τη πρόγραμμα και ποια είναι η αποτίμησή τη των επιστημονικών στοιχείων από πολλέ μελέτε που δείχνουν ότι οι ανιχνευτέ ψεύδους δεν είναι ε, ακριβεί. Επίσης, τι γίνεται με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων ερωτώνται με το σύστημα αυτό. Και τι γίνεται με τα προσωπικά του δεδομένα, όπω τι απαντήσει στι ερωτήσει που συλλέγονται. Και τρίτη και τελευταία ερώτηση, ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τα άτομα που ε, υποβάλλουν αίτηση για άσυλο στα σύνορα και τι δικαιώματα ή ένδικα μέσα του διατίθενται εφόσον ε, απομακρύνονται στα, στα σύνορα, διότι οι συνοριοφύλακε έλαβαν κάποια απόφαση αρνητική βάσει του ανεχνευτού ψεύδου. Ευχαριστούμε, Γιούντιθ. Οπότε, ε, επιπλέον ερωτήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε, Επιτροπή, σε τι ερωτήσει είστε θέση να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ ενώπιον των μελών της Επιτροπής σας για να μπορέσω να απαντήσω και να διευκρινίσω αυτά που ρωτήσατε για το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτούμε. Ε, να περάσω απευθείας στο δεύτερο τμήμα των ερωτήσεων αφού τονίσω ότι εδώ θέλουμε να απαντήσουμε μία από τις δύο ερωτήσεις που είχαν τεθεί εκ των προτέρων. Βεβαίω, όλες αφορούν το ίδιο θέμα, το ίδιο πρόγραμμα, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να απαντήσω σε όλα, εάν γίνεται. Ξεκινώντας, να πω ότι η Επιτροπή απάντησε πριν από λίγες μέρες στο Κοινοβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου ως προς την πρώτη ερώτηση Πολλά στοιχεία της απάντησής μας ήδη καλύπτονται στην ίδια την επίσημη απάντηση που αποβάλαμε. Πρώτον, λοιπόν, μιλάμε για έρευνα σε αυτό το πεδίο. Η έρευνα είναι ένα από τα στοιχεία που συλλέγονται ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση των συνόρων που είναι προτεραιότητα βεβαίως για μας. Άρα επενδύουμε στην έρευνα για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνολική διαδικασία του ελέγχου των συνόρων. Για το ίδιο το πρόγραμμα και αυτά που κάνει. Πρέπει να κάνω εδώ μια διευκρίνηση ευθύ αμέσω. Το πρόγραμμα δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία ενό συστήματο, την επιχειρησιακή του χρήση δηλαδή. Αλλά θέλουμε να δούμε κατά πόσον συγκεκριμένα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να είναι χρήσιμα στη διαχείριση των συνόρων και τη φύλαξή τους. Άρα το πρόγραμμα κοιτάζει μια σειρά από πράγματα, όχι απλώς να χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα ανείχνευση ψεύδου καλά και ντε. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να ελεγχθεί το κατά πόσον τα έγγραφα είναι αυθεντικά ή τα βιομητρικά δεδομένα ή ο εντοπισμός ε, παράνομων προϊόντων ή το κατά πόσον κάποιοι έχουν ε, αναζητήσει καταφύγιο σε κοντέινερ καθώς διασχίζουν τα σύνορα και ούτω καθεξής. Άρα ο σκοπός δεν είναι να εντοπίσουμε απλώς ενδεχόμενα ψεύδι στην αφήγηση κάποιου. Είναι ένα μέρος της προσέγγισης μας αυτό. Κάτι άλλο που κάνουμε, και αυτό αφορά όλες τις παραμέτρους του προγράμματος, είναι να κοιτάξουμε κατά πόσον ένα τεχνολογικό εργαλείο θα ε, είχε νόημα να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο ε, πλαίσιο. Δηλαδή, το θέμα του προγραμματός είναι να δούμε αν λειτουργεί καλά ή όχι, τι αποτελέσματα δίνει, βάσει επιστημονικών δεδομένων που συλλέγονται από την ίδια τη λειτουργία του προγράμματος. Εφόσον λοιπόν το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν είμαστε σε θέση να πούμε εάν η τεχνολογία επηρεάζει το αποτέλεσμα ή όχι. Αυτό θα φανεί αργότερα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα είναι ότι απλώς κοιτάζουμε αν έχει νόημα να μιλάμε για το θέμα αυτό από επιστημονική σκοπιά. Έχει νόημα να χρησιμοποιούμε κάποια τεχνολογικά εργαλεία σε συγκεκριμένου ε, τομεί, όπω η διαχείριση των συνόρων. Έπειτα, θα πρέπει να μελετήσουμε σε επίπεδο χάραξη πολιτική και λήψη αποφάσεων εάν θα ήταν καλό η τεχνολογία που έχει δοκιμαστεί ήδη να χρησιμοποιηθεί και να εξελιχθεί σε ένα επίσημο ε, πραγματικό εργαλείο για τους συνοριοφύλακες. Αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. Τώρα, όταν μιλάμε για τα δικαιώματα, τα ηθικά και θεμελιώδη δικαιώματα, διαβεβαιώ τα μέλη της Επιτροπής σας ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα κράτη-μέλη το ίδιο, ε, δίνουμε ύψιστη προτεραιότητα στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκδήλωση όλων αυτών των διαδικασιών και ιδίω στην έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε έρευνα που κάνουμε πρέπει να σέβεται τι παγιωμένε ηθικέ αρχέ και την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε ε, βήμα του προγράμματος έχει να κάνει με, το, με την ηθική σάρωση όπως λέγεται. Δηλαδή η ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περνάνε από κάθε στάδιο της διαδικασίας ε, και το περνάνε από την Κρυσάρα για να δούνε κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια του προγράμματος. Και μετά υποβάλλονται συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχει κάποιον έναν σύμβουλο για τα θέματα ηθικής που ασχολείται ακριβώς με το πρόγραμμα αυτό και μόνο και παρακολουθεί το πώς λειτουργεί σε όλες τις φάσεις, δίνοντας τις απαραίτητες συστάσεις και εντοπίζει τις κόκκινες γραμμές που δεν θα πρέπει να ξεπερνιόνται. Οπότε, ως προς την αξιολόγηση της ίδιας της πρότασης, θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι η πρόταση υποβλήθηκε για αποτίμηση από εξωτερικούς αναλυτές, οι οποίοι ανέλησαν από επιστημονική σκοπιά εάν η πρόταση αυτή καθεαυτή είχε τη δυνατότητα να μας δώσει κάποια αποτελέσματα. Και έτσι λήφθηκε η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με την πρόταση αυτή. Ε, ήταν από αυτές που είχε ε, συνεξεταστεί η πλέον πολλά υποσχόμενοι. Αυτή που υποσχόταν τα περισσότερα. Ε, επί των λεπτομεριών. Εδώ δεν μιλάμε για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για το σύστημα της ηλεκτρονικής διαχείρισης των συνόρων και αυτομάτως να βλέπουμε στο σημείο εισόδου ποιος πρέπει να μπει και ποιος όχι. Μιλάμε απλώς για την χρήση τεχνολογικών μέσων και το κατά πόσον αυτά εξυπηρετούν το σκοπό τους. Τώρα, εάν τα τεχνολογικά μέσα κρυθούν κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού και αν υπάρξει απόφαση να παραταθεί η χρήση τους και να ερευνήσουμε περαιτέρω τη χρήση των εργαλείων αυτών από τους συνοφυλακές, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θα κοιτάξει τη διαλειτουργικότητα των όσων ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισαγωγή ενός συστήματος αμοιβών δεν είναι μέρος του πεδίου του προγράμματός μας. Άλλα θέματα που θα μπορούσα να αναφέρω Όχι, νομίζω ότι θα πάψω. Θα πάψω εδώ. Θα απαντήσω όμως ευχαρίστως οποιασδήποτε επερωτήσεις της Επιτροπής σας. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι βεβαία ότι θα υπάρχουν επερωτήσεις. Εγώ έχω ήδη μία έτοιμη, αλλά πρώτα απ' όλα λόγω στη Σόφη. Πραγματικά πάντοτε αγχώνομαι. Όταν έρχεται εδώ ένας άνθρωπος με τις καλύτερες υποθέσεις του κόσμου, δεν έχω να πω, αλλά παρασύρεται από κάτι που είναι τόσο ανησυχητικό για τη δημοκρατία μας και κάθεστε εδώ και μας λέτε Κάτι που δεν βγάζει νόημα για μένα. Μα λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό γιατί έχει το μεγαλύτερο δυναμικό ε, να πετύχει του στόχου μα. Μα το νόημα, το ερώτημα είναι ότι ο βαθμό ακρίβεια είναι 76%. Αυτό το λέτε το μεγαλύτερο δυναμικό επίτευξη στόχων. Ε, τι ήταν τα άλλα προγράμματα δηλαδή. Και κάτι που πραγματικά εμένα με ε, κάνει να ε, έχω ζαλάδες είναι γιατί διαλέξατε την Ουγγαρία από όλα τα κατημέλη. Την Ουγγαρία μα προς Θεού. Και μετά λέτε ότι το σύστημα αμοιβών δεν είναι μέρος του προγράμματος. Ωραία. Αλλά στον ιστότοπο του συστήματος ε, του ηλεκτρονικού ελέγχου αναφέρεται. Και εάν δοκιμάζετε το σύστημα αυτό, γιατί δεν το δοκιμάζετε στον κύριο Τραμπ, εάν σας δώσει 100% ε, βαθμό ψεύδους, θα ξέρετε ότι λειτουργεί. Ότι δεν λειτουργεί. Ε, ευχαριστούμε η κυρία Βρεζιά. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, Σοφία για την ερώτησή της. και την Γιούντιθ, η οποία την επόμενη μέρα έθεσε μια παρόμοια. Συμμερίζομαι όλα όσα είπαν οι δύο συναδελφοί μου. Εγώ παρακολουθώ τα θέματα αυτά, νομίζω από τότε πρώτα εξελέγει Ευρωβουλευτής, δεν θυμάμαι τώρα ποιες ήταν οι πρώτες μας συζητήσεις με την Ενίσα, αλλά θυμάμαι τη δουλειά είχε προηγηθεί, συμμετείχα και τότε και όπως είπε η Σόφη, Είναι πρωταπριλιά άραγε. Εγώ ε, αναρωτιέμαι πώς βρισκόμαστε σε καμιά αμερικανική σειρά το Light to Me. Και θα θυμίσω τον. Ε, μήπως, και θα πω πώ έχει προσληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Τιμ Ροθ, ε, ο ηθοποιό. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων σα ασχολείται με την τεχνητή ευθεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει. Εκεί συμμετέχουν το Skype, η Bayer, η Airbus, η Bosch και η Orange, μεταξύ άλλων. Διερωτώ με λοιπόν πόσο ανεξάρτητα είναι όλα αυτά. Αυτοί οι εμπειρογνώμονε τι εξαρτησία έχουν σε σχέση με τα προγράμματα που προτείνονται. Εγώ έχω παρακολουθήσει όλα τα σχετικά προγράμματα για τον έλεγχο και την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Τη διαλειτουργικότητα την ψάχνουμε. Αυτό είναι ο στόχο. Είναι το στέγαστρο όλου του προγράμματο. Ο αριθμό εκατομμυρίων που έχει ε, αφιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη για να δημιουργήσει τεχνητά τείχη σε όλο το μήκο των συνόρων μα είναι τρομακτικό. Και έχω πάει στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας. Έχω πάει και είδα πώς λειτουργούν τα συστήματα που σκοπό έχουν να εντοπίσουν οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία, ακόμη και μέσα σε φορτηγά, σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Πραγματικά διαρωτώ με τι κάνουν αυτοί οι ανιχνευτέ ψεύδου. Τι παραπάνω θα μα πούνε, ε? Μόνο θα πουλήσουμε πάλι κι άλλο συστήματα υποτίθεται ασφαλείας, τα οποία δεν χρησιμοποιούν σε τίποτα. Μόνο θα ε, κάνουν ορισμένες πολυεθνικές να πλουτίσουν κι άλλο. Είναι λε και είμαστε σε καμιά φάρσο κομμωδία εδώ πέρα. Έτσι. Τι είναι ενιχνευτέ ψεύδου με όλα τα συστήματα που ήδη έχουν ε, εκτεπλωθεί και χρησιμοποιηθεί. Ποιον δουλεύετε, δουλεύετε ποιον. Δεν υπάρχουν πια, λέω, για ένα σημείο και μετά. Μιλάμε 4,5 εκατομμύρια για ποιο πράγμα. Για το τίποτα. Τι ακριβώ θέλετε να μα πείτε. Ε, θα συμφωνήσω απολύτως με τη Σόφη. Έχει δοκιμαστεί και μετά ε, λέτε ότι κάνατε τις πρώτες δοκιμές στην Ουγγαρία. Ε, τι λέτε για να έχετε τις καλύτερες δυνατέ, την καλύτερη δυνατή δειγματοληψία με τους συνηροφύλακες της Ουγγαρίας. Τι, τι να πω. Ε, αυτοί που μας ανησυχούν περισσότερο είναι ακριβώς οι Ούγγροι. Και νομίζω ότι εδώ πραγματικά βρισκόμαστε στα όρια του γελίου στην απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επίσημη, την οποία τη διάβασα προσεκτικότατα, είναι κλασική. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ε, ηθική και τα διοντολογικά, όλοι οι εμπειρογνώμονες τα σέβονται. Τι μα λέτε, αν θέλετε να είστε αξιόπιστοι, δώστε μα τα αποτελέσματα, αυτό που είπαν οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε λίγο να προχωρήσουμε και να έχουμε μια ελάχιστη αξιοπιστία. Διότι εγώ δεν μπορώ να πω κουβέντα, δηλαδή τι να πω όταν με ρωτάνε για τέτοια πράγματα για τη χρήση αυτού του, την εκτέλεση τέτοιου είδου κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επαναλαμβάνω, έχουμε ξεπεράσει τα όρια του γελίου. Ευχαριστώ πολύ. Προτού δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά για ε, απαντήσεις, θα ήθελα να προσθέσω κάποιες ε, εύκολες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα για να επιδιώξουμε το στόχο. Ποιο στόχο? Αναρωτιέμαι, αν διαβάσει κανεί την επίσημη απάντηση, ουσιαστικά είναι σαν να αυξάνεται την αποδοτικότητα. Πιανού και για ποιον. Και ποιο είναι αυτό ο σκοπό που υποκρύπτεται εδώ. Εάν δούμε την κατάσταση στα σύνορα, διαφορετικοί άνθρωποι πλησιάζουν τα σύνορα. Αλλά αν κάποιο ζητά προστασία, ο καλύτερο τρόπο να τον υποδεχτεί κανεί είναι με ένα μηχάνημα που θα αποφασίζει εκείνο αν πρέπει να μπει ή όχι και αν πραγματικά χρειάζεται προστασία. Δεν είναι μάλλον η δουλειά ενός συνολοφύλακα να λάβει την απόφαση. Εάν ζητά κανείς προστασία πρέπει να ενημερώνουμε αυτού που εργάζονται στο σύστημα ασύλου. Εάν κάποιος φέρεται εγκληματία, να ζητήσουμε από την αστυνομία να κοιτάξει τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά, είναι πολλά τα ερωτηματικά, αλλά γιατί διαλέξατε την Ουγγαρία. Ίσως, λέω εγώ, μπορεί να μας πείτε κάτι άλλο, τα κράτη-μέλη δεν ήταν έτοιμα να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί καταλαβαίναν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και σε ό,τι αφορά το χρήμα, ε, είναι ενδιαφέρον ότι με τις τεχνικές λύσεις πάντοτε καταφέρουμε να βρούμε κονδύλια. Όταν όμως μιλάμε για άλλα θέματα που χρειάζονται χρηματοδότηση, όπως την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ίδιων των ανθρώπων, τότε τα χρήματα μας λείπουν. Αυτό ήταν πολιτική τοποθέτηση και δεν ήταν ερώτηση για σας. Έχω μια επερώτηση από τη Ρομπέρτα Μετσόλα και ίσως και από τη Γιούντιθ Σαρχεντίνη. Ρομπέρτα, ευχαριστώ Πρόεδρε, με συγχωρείτε που άργησα. Άκουσα τη Σόφη και την Μαρία Κριστίν και τη Γιούντιθ και κοίταξα λίγο τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα και θέλω να προσθέσω στις ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν. Το εξής κάτι πληροφορίες ε, θα ήθελα σε σχέση με όσα βλέπω μπροστά μου. Αν καταλαβαίνω καλά, το πρόγραμμα αυτό θα λήξει τον Αύγουστο φέτο. Και μια σειρά από κράτη-μέλη που συμμετείχαν ε, πέρασαν από διαγωνισμό, εάν καλά κατάλαβα. Βλέπω, ας πούμε, ότι και η συνοροφυλακή της Λετωνίας συμμετέχει κάποια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Βασιλείου, κάποια από την Πολωνία, και από ένα ερευνητικό διαστημικό κέντρο στην Ισπανία κάποιοι. Ε, έχετε τίποτα πληροφορίες για το... Για ποιο λόγο πήγε εκεί που πήγε το πρόγραμμα αυτό. Και όταν ε, μαζέψετε αυτές τις πληροφορίες που λέτε για την προστασία των δεδομένων που λέτε ότι σέβεστε κτλ. κτλ. Υπάρχει το ερώτημα του τι θα γίνει με τις πληροφορίες αφού φύγουν από τους συνεροφύλακες. Σε ποια φάση, εάν προβλέπετε αυτό, γίνεται ανάλυση των πληροφοριών σε συνδυασμό με την αίτηση ασύλου, τη διαδικασία δηλαδή εξέταση τη αίτηση ασύλου, αν κάποιο υποβάλλει αίτηση ε, διεθνού προστασία, αυτό εξετάζεται μετά τον αυτόματο έλεγχο ταυτόχρονα και μέσα σε τι χρονικό περιθώριο. Διότι αν λέμε ότι είναι αποτελεσματικότερη διαχείριση και ο έλεγχος των συνέρων, τι αριθμούς έχουμε για τι αιτήσει που απορρίπτονται και αυτέ που δεν απορρίπτονται και για όσου ε, γίνονται δεκτοί και όσου όχι. Ευχαριστούμε, Γιούντι Αρχεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ερωτήσει που προσέθεσα σε αυτέ τη σόφη δεν απαντήθηκαν. Περιμένω γραπτέ απαντήσει και βεβαίω η δική μου προθεσμία έχει λήξει πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να επαναφέρω τι ερωτήσει μου στην ημερησία διάταξη τη ΛΥΜΠ αργότερα, αλλά θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση επίσημη. Και επίση αυτό που θέλω να καταλάβω, όταν κονδύλια ξοδεύονται για την έρευνα, η απόφαση τη εκτέλεση των κονδυλίων δεν γίνεται μόνο στο επίπεδο των τεχνικών θεμάτων. Θα πρέπει κάτι να σα απασχόλησε και ω προ την ηθική και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και ακόμη και αν πέτυχε 100% το σύστημά σας, θα θέλατε να εφαρμοστεί στην Ένωση και να χρησιμοποιηθεί. Το ερώτημα αυτό σας έχει απασχολήσει καθόλου, έχει απαντηθεί. Διότι αν δεν σας έχει απασχολήσει καν, νομίζω, δεν θα έπρεπε να είχατε ξοδέψει όλα αυτά τα ε, ποσά. Και εάν είχατε κάποια απάντηση στο ερώτημα, καλό θα ήταν να τη μοιραστείτε και μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα να επιστρέψουμε στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αν και μεταξύ τους κάποιες ταυτίζονται φαίνεται. Προσπαθώ λοιπόν να τις ε, συνδυάσω όπου δυνατόν. Καταρχάς, στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα και ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι. Όχι. Εν τέλει το σχέδιο αυτό θα δώσει τα επιστημονικά δεδομένα που θα μας πούν αν δουλεύει ή όχι τεχνολογία αυτή. Θα στηρίζονται λοιπόν σε έναν αριθμό επιστημονικών μελετών που έχουν ε, διεξαχθεί σε κλειστό περιβάλλον και που δείχνουν πως αυτή η τεχνολογία μπορεί σε λειτουργικό περιβάλλον να φέρει αποτελέσματα, όχι όμως σε κάθε μορφή διάγνωσης ψεύδους. Για την ε, στόχευση αυτού του προγράμματος, λοιπόν, μόνο στο τέλος μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία. για την δυνατότητα χρήση σε λειτουργικό περιβάλλον ε, αυτής της τεχνολογίας και αυτά όλα, γιατί πρόκειται βέβαια για έρευνα. Η έρευνα μας δίνει μια δυνατότητα να κατανοήσουμε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να ισχύει. Και μετά μόνο τίφτε το θέμα και είναι όντως πολιτική επιλογή. Η απόφαση για την χρήση τεχνολογίας αυτής. Γιατί στην ε, Ουγγαρία. Κοιτάξτε, δεν αποφάσισε η Επιτροπή. Δεν αποφασίζει η Επιτροπή αν πρόκειται να γίνουν πιλωτικά σχέδια. Κατατίθενται προτάσεις από συμπράξεις με, πρωτα... ιδέες για το πώς θα γίνει αυτή η ερευνητική δραστηριότητα και εν τέλει αποφασίζουμε εάν θα δεχθούμε ή όχι. Και αυτό από ανεξάρτητους φορείς, όχι από την Επιτροπή την ίδια. Έτσι, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στη σύνθεση των συμπράξεων και να πούμε «Α, έπρεπε να είναι αυτό το κομμάτι έτσι ο ένας εταίρος να μην υπήρχε, ή να υπήρχε ένας άλλος. Όχι. Τεχνητή νοημοσύνη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων εγκαθιδρύθηκε το 2018 μετά την εκκίνηση του προγράμματος, άρα δεν μπορούσαν να έχουν συμμετάσχει σε κάποια αξιολόγηση αποφάσεων για την εκκίνηση των προγραμμάτων. ως προς την ουσία της σύνθεσης δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητήσουμε την αξία των ίδιων των εμπειρογνωμόνων. Χρήματα, ναι, πολλά χρήματα σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Ίσως μάλιστα κάποια αναφέρεται πως ε, αγγίζουν ε, παρόμοιους τομείς ή έχουν μια επικάλυψη. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό παρέτα είναι αρνητικό. αφενός με να έχουμε μια τεχνολογία, μια λύση που προτείνεται, μπορούμε, χάρη στην πολλαπλή αυτή έρευνα, να έχουμε εξέταση δυνατοτήτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και διάφορες ε, λύσεις πολιτικές ή άλλες με βάση αυτά. Και από την άλλη, Πάντα κοιτάμε και διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Μπορεί να έχουμε δηλαδή μια απόφαση ή, εν πάση περιπτώσει, ε, σε αφηρημένους όρους να συζητήσουμε τη δυνατότητα να αναστήσουμε ένα εργαλείο που είναι διαθέσιμο στην αγορά. Αυτό είναι πάλι μια απόφαση πολιτικής. Ή μπορεί να επιλέξουμε ε, να αναζητήσουμε νέε δυνατότητες για μια προσεχή γενιά Δηλαδή να πούμε ότι ξεκινάμε με, με αυτή τη διαθέσιμη τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουμε να βρούμε λύσεις και για το μέλλον και άρα στρεφόμαστε προς ε, συστήματα νέας γενιάς, τεχνολογία νέας γενιάς. Αντί να αντιδρούμε δηλαδή σε μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ και τώρα, να αναζητούμε και για το μέλλον προοπτικές. Αυτό πάντα ισχύει για την έρευνα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ε, τεχνολογία που θα είναι διαθέσιμη να χρησιμοποιηθεί από αύριο το πρωί, ο, ο κύκλος της, της έρευνας είναι μακρύς. Μέχρι και 7-8 χρόνια μπορεί να πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη το, την προέλευση των αιτημάτων. και το λόγο. Δηλαδή, αν ο κλάδο ο ίδιο ζητεί κάτι καινούριο, πώ είναι μόνο και μόνο για να αποκομίσει κέρδο. Εμεί βέβαια θα πρέπει αυτό να προσπαθούμε να το αποφύγουμε, αν ισχύει. Στον ορίζοντα 2020 που βλέπουμε τώρα σε εξέλιξη, ακριβώς κοιτούμε την ε, αναγνώριση των αναγκών του τελικού χρήστη, δηλαδή στόχος έρευνας που συζητείται διεξοδικά με τα κράτη-μέλη στην Προγραμματική Επιτροπή και ε, αιτήματα που πρέπει, τα αιτήματα για την έρευνα δηλαδή, να προέρχονται αλλά και τα λειτουργικά, από εκείνους που κάνουν τη δουλειά, που ασχολούνται με το θέμα αυτό καθημερινά. Εάν αρχική, το αρχικό αίτημα που οδηγεί στη περίληψη μιας ιδέας στο πρόγραμμά μας προέρχεται από τελικό χρήστη, προσπαθούμε να κοιτάξουμε και την ε, υποχρεωτική συμμετοχή των οργανώσεων των τελικών χρηστών στα προγράμματα, να την εισαγάγουμε, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οτιδήποτε ε, προτείνεται αντιστοιχεί όντως στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Και αυτό και γιατί πιστεύουμε ότι είναι η σωστή προσέγγιση αυτή. διοντολογία. συστάσεις βεβαίως είναι συστάσεις που συμμερίζεται και η Επιτροπή με βάση και τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούν και τα κράτη-μέλη. Και με την ε, ε ανάθεση σε έναν ε, η Θεωρητή Δεοντολογίας, η Σύμβουλο Δεοντολογίας. Μετά, στο ερώτημα αν θέλουμε μια μηχανή να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό μας. Εκεί θα απαντήσω ευθέως όχι. Ούτε καν είναι αυτή η επιλογή μας ή ο δρόμος που έχουμε πάρει. Άλλωστε είναι ήδη μέσα στο πρόγραμμα το ίδιο. Η ιδέα πως παραμένει πάντα ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Το μηχάνημα δηλαδή μόνο υποστηρίζει τον τρόπο λήψη αποφάσεων, προσφέρει τα στοιχεία που θα διευκολύνουν, αλλά δεν αποφασίζει το μηχάνημα. Την τελική απόφαση δεν παίρνει το μηχάνημα. Βοηθεί όμως τον συνοριοφύλακα να κάνει κάποιες εκτιμήσεις, τον ε, αφυπνίζει, εάν χρειάζεται, ε, σε ένα ζήτημα ιδιαίτερη ευαισθησία. Πάντω δεν αντικαθιστά τον συνοριοφύλακα ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Η γραμμή του χρόνου για το άσυλο δεν μπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, πεδίο δράση του προγράμματος. Το πρόγραμμα σας στόχο έχει να εξετάζει την αποτελεσματικότητα ορισμένων προγραμμάτων στην αντιμετώπιση ε, συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν οι τελικοί χρήστες εντοπίσει. Πώς τώρα αυτή η τεχνολογία μπορεί να οδηγεί στη λήψη κάποιων συγκεκριμένων αποφάσεων ή σε ποια χρονική στιγμή ε, μπορεί να παρέμβει η τεχνολογία ή σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι αξιόπιστη η τεχνολογία, πώς ε, συνδέεται με άλλα θέματα, ε, απαντήσεις σε προβλήματα για τους αισθούντες άσυλο κτλ. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να καλυφθεί σε όρους πολιτικών μελημάτων. εάν ναι, θέλουμε να δούμε το τελικό, τελική έκβαση σε αυτούς τους όρους. Ε, νομίζω ότι έχω ήδη δώσει απαντήσεις σε όλες τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας θυμίζω ότι ήδη έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Εκμεταλλευόμαστε βέβαια το γεγονός ότι ξεκινήσαμε πολύ νωρίτερα τη συζήτηση του θέματος αυτού. Σας θυμίζω όμως ότι ήδη έχουμε εξαντλήσει το θέμα αυτό. Δίνω ωστόσο το λόγο για άλλη μια φορά στην ε, Σοφίν Φέλντ, εφόσον την ενδιαφέρει. Για να συνεχίσει, αλλά σας υπενθυμίζω ότι Η παρουσία του εκπροσώπου τη επιτροπή εδώ οφείλεται στο ότι έχει να παρουσιάσει το ερευνητικό αυτό θέμα και όχι ότι πρέπει να συζητηθεί κάθε πιθανό ζήτημα. Κυρία Νιφέλτ. Ναι, θα επαναλάβω αυτά που έχω επαναλημμένως πει. Πιστεύω και επιμένω ότι θα πρέπει ο, ή, ο ίδιος ή η ίδια η Επίτροπος να έρθει να δώσει απαντήσεις. Και χωρίς να θέλω να διατυπώσω καμιά προσωπική αιχμή. Είναι ζητήματα πολιτικά αυτά και κάθε φορά είναι ανεπαρκείς οι απαντήσεις που μας δίνονται. Και για μας και για την ε, Επιτροπή μας. Δεν μπορεί να έρχεται η Επιτροπή να μας δίνει τέτοιες γραφειοκρατικές απαντήσεις και να μας ξαποστέλνει σαν να είμαστε παιδιά του νηπιαγωγείου. Έχουμε να δώσουμε λογαριασμό στους πολίτες. Ε, είναι παράδεκτη κατάσταση. Και επίσης, έτοιμα για πρόσβαση στα έγγραφα. Έχω διατυπώσει, Διαρκώ αναβάλει την ε, πρόσβαση η Επιτροπή, χρειάζονται απαντήσει, ειδικά με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Έχουμε εκπροσώπους του κλάδου με άμεσο συμφέρον. Έτσι όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις για την ε, χορήγηση κονδυλίων πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα στα όλα τα έργα, όλα τα σχέδια. Και όχι να μας λέτε του χρόνου. Ευχαριστώ. Καλώς. Άρα δεν ήταν πρόσθετη η ερώτηση αυτή. Ε, συμφωνώ ωστόσο πως υπάρχουν εκκρεμότητες και εν γέννη ζητήματα ανοιχτά Οι εμπειρογνωμόνες ούτως ή άλλως από τον κλάδο προέρχονται και ο τελικός τους στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Βεβαίω και πρέπει μια μελέτη να απευθύνεται στον τελικό χρήστη, αλλά εδώ ο τελικό χρήστη είναι οι συνοριοφύλακε. Σε άλλε, ε, πολλοί άλλοι όμω είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συναφή δράση. Δεν μιλάμε δηλαδή για τον έλεγχο για τους πολίτες, τους μετανάστες ή τους ετούντες άσυλο. Επομένως η αναφορά στον τελικό χρήστη δεν αρκεί νομίζω. Και γι' αυτό χρειάζεται η επαλήθευση ανθρωπινών δικαιωμάτων στο τέλος αυτής της ε, μελέτης. με ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ευχαριστώ τους συναδέλφους λοιπόν που είναι εδώ, που περίμεναν και διατύπωσαν τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ την Επιτροπή που έδωσε τις απαντήσεις. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Μην ξεχνάτε όμως ότι αύριο το πρωί έχουμε ακόμα μια συνεδρίαση Επιτροπής μας. 9 το πρωί. Ευχαριστώ.